Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. E, Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα. θα πρέπει να έχετε λάβει την ε, ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδριάσους, Προβαίνουμε τώρα στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας υπενθυμίσω σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε το αρχικό ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής ε, συνεδριάσεως υπάρχει διερμηνία από και προς τις γλώσσες που χρησιμοποιούν τα πλήρη μέλη της υποεπιτροπής μας Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Εκτός αν υπάρχουν κάποιες ε, παρατηρήσεις και σχόλια, θα θεωρήσω ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Επίσης θα έχετε λάβει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Υποεπιτροπής μας, της συνεδριάσεως μάλλον, της 24 η Σεπτεμβρίου και της 13ης Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος ε, του απογεύματος σήμερα, θα θεωρηθούν τα πρακτικά ως εγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε και να πάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο, ο πρεσβευτής, ο κ. Walter Stevens, που είναι πρόεδρος του PSC, για εκείνους από εσά κυρίες και κύριοι που είσαστε από παλιά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και μέλη εδώ της Επιτροπής για την Ασφάλεια θα τα γνωρίζετε καλά υπό την παρούσα του ιδιότητα και θα το γνωρίζετε και από προηγούμενες ιδιότητες ε, ήταν προσκεκλημένο σε συνεδριάσεις μας και είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει για το πλαίσιο της ΚΕΠΑ το τοπίο που μεταβάλλεται της ασφαλείας και ελπίζω και για όλες τις σχετικές διαδικασίες θα μας ενημερώσει λοιπόν για τις τρέχουσες προκλήσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις του PSE. Κύριε Πρεσβευτά, κύριε Στίβενς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και δικαιωμένα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε που είχα την καλοσύνη να με καλέσετε σε αυτή τη διακεκριμένη υποεπιτροπή. Σχεδόν ένας χρόνος πέρασε από όταν είχα ξαναέρθει στην Επιτροπή 27 Νοεμβρίου με την πρώτερη σύνθεσή της, σχεδόν ένα χρόνο πριν. Πολλά έχουν αλλάξει και βέβαια και στη γειτονιά μας έχουν αλλάξει πολλά αλλά και στην Επιτροπή, διότι βλέπω αρκετά καινούργια πρόσωπα, αλλά και κάποια αρκετά γνωστά. Θέλω να τονίσω εξ αρχής ότι θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί σας για να εξετάζουμε τα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας και θέλουμε να είμαστε πιο ορατοί, πιο αποτελεσματικοί και να έχουμε και μεγαλύτερη επιτόπου επιρροή. Μου ζητήσατε να μιλήσω για τις προτεραιότητες της ΚΕΠΑ στα πλαίσια της μεταβαλλόμενης ε, ατμόσφαιρας στον τομέα αυτό της ε, ασφαλείας και οι μεταβολές είναι τάχιστες, το περιβάλλον μεταβάλλεται τάχιστα και είναι κάτι που πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμεθα. Θα ξεκινήσω, εφόσον είστε πολύ καινούργοι, ότι και ΠΑ βασίζεται επί τριών πυλώνων. Ο ένας είναι επιχειρήσεις, το άλλο είναι δυναμικό δυνατότητες και το άλλο είναι συμπράξεις, εταιρικές σχέσεις. Είναι προτεραιότητες όλες αυτές και σχετίζονται με αυτά που το Δεκέμβριο του 2013 έθεσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ως προτεραιότητες. Όσον αφορά επιχειρήσεις, έχουν πέντε θετικές επιχειρήσεις για την ώρα και 11 πολιτικές. Η πλέον επιτυχής είναι η επιχειρήση κατά των πειρατών Αταλάντα, Ιούφορ, Αταλάντη και έχουμε και μια νέα πολιτική αποστολή στο Μαλί Τώρα το δυναμικό μας, οι δυνατότητές μας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να παρέχει ασφάλεια. Και αν θέλουμε αυτό χρειάζεται να υπάρχει το δυναμικό. Και ε, δεν έχουμε δυνατότητες σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν ε, το προσωπικό, το δυναμικό και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και περιπλέκονται τα πράγματα και μειώνονται και οι προπολογισμοί ε, και προσπαθούμε να κάνουμε επιμερισμό και διαμοιρασμό των διαφόρων δυνάμεων που έχουν τα κράτη-μέλη και θέλουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες εκεί που μας λείπουν, όπως τη Λιβύη, όπου μας έλειπαν οι δυνατότητες όπως ο νεφοδιασμός, ε, ο εναέριος και τα drones ή τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη ή συστήματα και θέλουμε να έχουμε και τη σωστή βιομηχανική βάση. Η Claude Fons ε, νομίζω ότι σας έχει εξηγήσει περαιτέρω το θέμα. Να σκιαγραφίσω την κατάσταση. Τάσεις που υπάρχουν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον βέβαια. Πρώτα απ' όλα έχουμε λοιπόν τη μεταστροφή, τη στροφή των ΙΠΑ προς την Ασία και αναμένεται εξ αυτού ότι η Ευρώπη θα απομειστεί περισσότερε ευθύνε για τη δική τη ασφάλεια. Το είδαμε και στη Λιβύη, το είδαμε και στο Μάλι, το βλέπουμε σε κάποιο βαθμό και στην ε, Ουκρανία. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει και κάποια αντίφαση αυτό. Και μια στιγμή όπου τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττονται από μια οικονομική κρίση. Και αισθάνεται κανείς ότι παντού στις συζητήσεις, στους διάφορους φορείς βλέπει κανείς ότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες και περιπλέκει τη ζωή μας. Ίσως σαν αποτέλεσμα αυτού, και αυτή είναι τρίτη τάση, βλέπουμε λοιπόν μια αύξηση ρεαλισμού έναντι της θεωρίας. Στην αρχή και πά αφορούσε περισσότερα σύμβολα, ε, θεωρίες, ε, αρχηγία, πριν βασική στόχη, στρατιωτικός τομέας, πολιτικός τομέας, 10.060 άνθρωποι διατίθεται για κάποιο σκοπό. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει σαν ανάλυση. Τα κράτη-μέλη κινούνται περισσότερο προς πραγματιστική προσέγγιση. Για το θέμα είναι τι μπορούμε να μπορούμε να ε, στείλουμε εκεί, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να ελεγχθεί η κατάσταση όπως στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Δεν λέω ότι αυτά τα θεωρητικά στοιχεία απομακρύνονται, αλλά επικρατεί κυρίως η πραγματιστική θεώρηση. Τέταρτον, κάτι σχετικό με το νέο περιβάλλον, τη μειώσεως των πόρων. Τονίζεται περισσότερο η ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή, ε, είναι πολύ σημαντικές οι αποστολές και επιχειρήσεις, αλλά είναι ένα στοιχείο της προσέγγισης, σημαντικό στοιχείο και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολιτική. Αποτελούν τμήματα ευρύτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης, χρειάζονται διπλωματικά μέσα, αναπτυξιακά μέσα, αλλά βέβαια και αμυντικά συστήματα και συστήματα ασφαλείας και αυτά χαρακτηρίζονται από μια νέα προσέγγιση που παρακολουθούμε, το βλέπουμε σε μια κρίση. Εκπονούμε ε, πλαίσιο πολιτικής για ανταπόκριση σε μια κρίση προσέγγιση για την κρίση. Προσπαθούμε να δούμε πιο σφαιρικά τις κρίσεις. Πέμπτον, ε, πολύ δύσκολο το ε, περιβάλλον, πιο επικίνδυνο, πιο περίπλοκο. Η συνεργασία με τέρους όλο και περισσότερο αποτελεί αναγκαιότητα. Και το βλέπουν να ξανά τάση και το ΝΑΤΟ βέβαια είναι αρκετά σημαντικό, αλλά και η Αφρικανική Ένωση, ο ΙΕ. Συζητούμε με τον ΙΕ τώρα πώς ε, πρέπει να προσέξουμε το θέμα. Το ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντικό. Χτες σε μια συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας, ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μίλησε για τις εταιρικέ σχέσεις, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Επίση, εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεω αυξάνεται η τάση για συμπράξει και εταιρικέ σχέσεις, διότι τα διάφορα μέσα και εργαλεία πρέπει να συναθριστούν και το προβλέπει και η Συνδική της και υπάρχει αυξανόμενη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπω εδώ εκπροσώπους αυτής σε μεταβατικές καταστάσεις Εφερρυπίν. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα αποτελέσματα αποστολών της ΚΕΠΑ μακροπρόθεσμα όταν αναλαμβάνουν μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά. Οπότε αυξάνεται η τάση για εταιρικέ σχέσεις Όμω όλα αυτά εκτιλήσονται ακόμα και περιμένουμε και πολλά από το νέο είπατε Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία εξωτερική δράση πρέπει να πλησιάσουν οι φορεί και τα μέσα, αλλά σημειώνεται πρόοδος. Και το βλέπω και τώρα και σε πρώτερες, όταν, ιδιότητες που είχα δύο περισσότερες άλλες τάσεις. Βλέπω ότι και στην ΚΕΠΑ υπάρχει μεγαλύτερη τάση προς την ανάπτυξη δυναμικού και σχετικές αποστολές και για το στοντικό τομέα και για τον πολιτικό τομέα ισχύει κάτι τέτοιο. Βλέπετε τι γίνεται στο Σαχέλ, στην Ουκρανία, τι προσπαθούμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε δυναμικό, να δώσουμε συμβουλές, να εκπαιδεύουμε ούτω ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους εταίρους μας, στις χώρες, να αναλάβουν στα χέρια του την ασφάλειά τους και αυτό ίσως είναι η τελευταία τάση που θα ήθελα να τονίσω. Ε, βέβαια πολλές από τις αποστολές μας εξακολουθούν να είναι στην Αφρική. Σίγουρα είναι το κέντρο βάρου των δράσεών μας. Ε, βλέπετε επίσης και μια τάση προς την ε, γειτονιά αποστολές στην Ουκρανία, ακόμα και με τρίο μεγέθους, Λιβύη, όπου έχουμε προβλήματα βέβαια, αλλά βλέπετε μια αλλαγή και εκεί. Βέβαια Αυτά είναι κάποιες γενικές τάσεις εγκάρσιες, αλλά υπάρχουν και κάποιες νέες προκλήσεις και προβλήματα και με τα προβλήματα έρχονται και ευκαιρίες. Η πρώτη πρόκληση, ευκαιρία, ας το πούμε ευκαιρία, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Άμυνα και την Ασφάλεια που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο που καθόρισε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα χρόνια και πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι πολύ σημαντικές στιγμές αυτές. Μέχρι τώρα συνεχίδαμε συνέχεια στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου άμενης και ασφαλείας, αλλά έχουμε νέα προθεσμία μπροστά μας, όπου είναι το Συμβούλιο του Ιουνίου. Και εκεί οι ηγέτες θα αποτιμήσουν τα όσα συνέβησαν από το Δεκέμβριο του 2013. Θα αυξηθεί η πίεση λοιπόν να επιτύχουμε αποτελέσματα. Και, ξ... και ε, θέλαμε να δώσουμε ορατότητα και να υπάρχει αποτελεσματικότητα των δράσεών μας. Ε, μετά χρειάζεται δυναμικό και τρίτον ε, χρειάζεται βιομηχανική βάση. Νομίζω ότι είπατε η αρμοστία ετοίμασε έκθεση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτευθύνσα πρόοδο. Εν γέννη όμως και οι Υπουργοί Άμυνας το Νοέμβριο σίγουρα θα τα συζητήσουν αυτό. Είναι σημαντική στιγμή θα τα λάβουν υπόψη όλα αυτά και τα προωθήσουν. Εν γέννη δεν είναι εύκολες οι συζητήσεις και η πρόοδος υπήρξε αρκετά αργή, δεν είναι κάτι εύκολο, βέβαια εξαρτάται κατά πολύ από τα κράτη-μέλη και βέβαια είναι πολύ δυσχερέ το περιβάλλον, παρότι θα ρωτούσε κανείς ότι η ομαδοποίηση, το pooling and sharing είναι μια φυσική προσέγγιση, αλλά υπάρχουν πολλοί όροι και πολλά εμπόδια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ε, δεν έχουμε ήδη κάποια αποτελέσματα όπως κυβερνοασφάλεια, αμυντική πολιτική στον κυβερνοχώρο, στρατηγική ασφάλεια στις θάλασσες και το σχέδιο δράσης. Είναι μια ευκαιρία αλλά και πρόβλημα να προχωρήσουμε και οι πιέσεις θα αυξάνονται για να προχωρήσουμε πάνω σε όλα αυτά. Κάτι σχετικό Κάτι που αντιμετωπίζει η Εξωτική Επιτροπή είναι η τέταρτη γενιά. Λοιπόν, ξεκινάμε τις αποστολές όπως στην Αφρικανική Δημοκρατία. Όλοι λένε ότι αυτό χρειάζεται διότι βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, σχεδόν μαζικές δολοφονίες και πρέπει κάτι να κάνουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινητοποιήσουμε επαρκείς ε, δυνάμεις. Επίσης αληθεύει και για τις πολιτικές αποστολές. Ε, και εκεί παίζει ρόλο το οικονομικό πλαίσιο και δημιουργεί προβλήματα. Η τέταρτη αυτή γενιά είναι ένα πρόβλημα. Επίσης άλλο θέμα είναι ο προπολογισμό. Και είναι ο προπολογισμό για την ΚΕΠΑ, όπου τώρα υπάρχει ένα ανώτατο όριο από φέτο, μια οροφή. Θα έλεγε βέβαια ότι σε περίοδου λιτότητα είναι συνηθισμένο να υπάρχουν ανώτατα όρια. Το πρόβλημα όμω το μεγάλο είναι μεταξύ των πιστώσεων, υποχρεώσεων και πληρωμών. Ε, ούτως ώστε να μπορέσεις να ξεκινήσεις ε, μια δράση αλλά το πρόβλημα είναι αν στο τέλος η πιστός πληρωμών είναι το μισό των αναλήψεων υποχρεώσεων ε, σταματάς. Δεν μπορείς να πληρώσεις αυτά που έχεις αναλάβει. Οπότε είναι μεγάλο πρόβλημα. Συζητείτε το θέμα στην Επιτροπή και στην Ρίλεξ. Θέλουμε να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε μια άλλη λύση, να βρούμε άλλες πηγές χρηματοδοτήσεως. Επίσης που μπορούμε να θέσουμε πώς μπορούμε να θέσουμε τις προτεραιότητες, τι μπορούμε να κάνουμε για οικονομίες, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα, ούτω ώστε να μειώσουμε το κόστος των αποστολών και καμιά φορά και το κόστος ασφαλείας που είναι πολύ ψηλό. Όταν έχουμε επιχειρήσει στο Αφγανιστάν ή στη Λιβύη δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανθρώπους μας εκεί ε, στο πεδίο χωρίς επιτόπου, χωρίς προστασία. Και μετά είναι οι δημοσιονομικές πτυχές της χρηματοδοτήσεως της ΚΕΠΑ για τα στρατιωτικό τομέα έχουμε το θέμα τη αναθεωρήσεως του μηχανισμού Αθηνά και υπάρχουν προτάσεις επιτάπητος που δυσκολεύουν κάποια κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει η αναθεώρηση του μηχανισμού Αθηνά για τη χρηματοδότηση. Πώς μπορούμε να τα θέσουμε στο κοινό κόστος. Ας στείλουμε μια ομάδα μάχης. Ε, το κόστος της μεταφοράς μπορεί ίσως να ενταχθεί στις κοινέ ταπάνες. Υπάρχουν και άλλα θέματα από την πολιτική πλευρά όπως το κέντρο κοινών υπηρεσιών, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συμπράξεις, συνέργειες οικονομικές συνέργειες μεταξύ στατιωτικών αποστολών και πολιτικών. Πρέπει να δούμε πράγματο χάρη πώ μπορούμε να έχουμε... Ε, στο Μαλί έχουμε την αποστολή και με την νέα πολιτική αποστολή μπορούμε να, να είναι στους, στον ίδιο χώρο όπως η στατιωτική αποστολή, να κατέχουν τον ίδιο χώρο μειώνει το κόστος αλλά έχει και κάποιες συνέπειες όσον αφορά τις ηγετικές δομές, αυτονομία επιχειρήσεων κλπ. Και τρίτο στοιχείο όσον αφορά το οικονομικό θέμα είναι οι δημοσιονομικοί κανονισμοί. Ανακαλύπτουμε και ανακαλύπτουμε συνεχώς ότι καμιά φορά δημοσιονομικοί κανονισμοί που βέβαια ε, αναφέρονται σε όλους τους κανόνες, στους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, πάντα ε, ασχολούνται, καλύπτουν τις περιπτώσεις κρίσεων, αλλά δεν ξέρω να πάντα με τον δεδειγμένο τρόπο. Τι είναι δυνατόν στην ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να δούμε ότι γίνονται γρήγορες εκταμιεύσεις, ταχεία δράση είναι δυνατή, αλλά δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό στον τομέα της διαχείρισης των κρίσεων και των σχετικών μέσων και αυτό κάπως παρεμποδίζει μια ταχεία αντίδραση. Είναι εξίσου σημαντικό και για τις στρατηγικές της μεταβατικές όπως αποκαλούνται. Έχουμε τις αποστολές και επιχειρήσεις και ΠΑ, στο Κονγκό παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν ε, ε, επιχειρήσεις που ασχολούνται με κρίσεις, όμως όταν μιλάμε για τον τομέα της ασφαλείας στο Κονγκό πολλοί άνθρωποι μένουν εκεί επί μακρόν. Οι άνθρωποι μας μένουν επί μακρόν χρονικό διάστημα. Και πρέπει να εξετάσουμε κάτι με τη μετάβαση. Να δούμε πώς γίνεται η μετάβαση. Πώς θα αλλάξει η αποστολή τη ΚΕΠΑ μέσω μακροπρόθεσμου εργαλείου, μέσω αναπτυξιακή συνεργασία. Οπότε είχαμε ένα-δύο καλά παραδείγματα. Το Κονγκό είναι ένα όσον αφορά την πολιτική πλευρά. Οπότε είχαμε την Ιούπολ και από τη πλευρά ε, για να δούμε πώς μπορούμε να, να αλλάξουμε την προσέγγιση της ΚΕΠΑ, να, να ξεφύγουμε, να ολοκληρωθεί η ΚΕΠΑ, η αποστολή ΚΕΠΑ και να διατηρηθούν, υπάρχει βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της αποστολής, να μην χάνονται και να αναλαμβάνονται από άλλα μέσα και εργαλεία. Μια άλλη πρόκληση είναι η υλοποίηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Υπάρχουν κάποια νέα πράγματα στη συνθήκη τη Λισαβόνα, όπω το άρθρο 44 που σημαίνει ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει εντολή σε μια ομάδα χωρών ή σε μία ή δύο χώρε να κάνουν κάποια πράγματα μέσα στο πλαίσιο μιας, της αντιμετώπισης μιας ε, κρίσης και μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας έχουμε και το, τα αντίστοιχα κονδύλια δεν υπήρξε όμως μεγάλη πρόοδος, υπήρξε πολλή συζήτηση αλλά όχι πρόοδος επειδή είναι διχασμένα τα κράτη-μέλη επ' αυτού. Αυτό που βλέπουμε φυσικά είναι η ανάγκη πολιτικών αποφάσεων γιατί όταν είναι διχασμένα τα κράτη-μέλη και έχουν διαφορετικές απόψεις είναι περίπλοκη υπόθεση. Είναι θέμα λοιπόν πολιτικής βούλησης και το θέμα του πώς θα μπορέσουμε με την εντολή να δράσουμε για την χρήση battle groups ε, όπως ε, στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Όπως είπαν ότι μπορούμε να αποστείλουμε μια τέτοια ομάδα στρατιωτική Ωστόσο δεν υπήρξε πολιτική συμφωνία, πολιτική βούληση να γίνει χρήση της ε, Bat Group των ενόπλων ομάδων ισχυματισμών εκεί. Όμως, Πρόεδρε, το, η μεγαλύτερη πρόκληση φυσικά είναι κάπως αυτό το απόλυτα νέο περιβάλλον, το νέο περιβάλλον ασφάλειας και το πώς αντιδρούμε σε αυτό. Και αυτό βρίσκεται επίσης στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να πω όταν συναντήθηκαν οι ηγέτες μας το Δεκέμβριο του 2013 ήδη είχαν αναγνωρίσει τις σημαντικές αλλαγές και τα όσα είχαν μεταβληθεί σε σχέση με το περιβάλλον ασφάλειας, με την αντιμετώπιση προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, δημοκρατίας, πάσης φύσεως φαινομένων και ο συνδυασμός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας στα θέματα. Αλλά και πάλι όταν συνήλθαν δεν, θα, μπορούσαν να φανταστούν ότι θα προσαρτούσε η Ρωσία την χερσόνησο της Κρυμαίας και ότι θα δημιουργούσε αυτό τεράστια πίεση από πλευράς και του ISIS, του Ισλαμικού κράτους για, την, για το Ιράκ και τη Συρία και με τις δράσεις του ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια τέτοια τεράστια απειλή και σε σχέση με την αντιμετώπιση της ε, αυτής της ε, ομάδας εξεπλάγησαν όλοι και είπα και αν δούμε την Ουκρανία και για την κατάσταση εκεί φυσικά έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα το πλαίσιο της ασφάλειας το τοπίο για την ασφάλεια στην Ευρώπη η αλλαγή συνόρων δια της βίας είναι κάτι απόλυτα απαράδεκτο και κάτι το οποίο παραβιάζει και παραβαίνει στις αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκη. Αυτά σε σχέση με την ενημέρωσή, ενημέρωσή σας. Να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια σημαντικότερα σημεία Διατηρήσαμε πολύ στενή συνεργασία, ενότητα με τόπου με τους διατλαντικούς εταίρους μας, συμμάχους μας και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και από πλευράς μας είχαμε δύο τέτοιες συναντήσεις όπου το συμπέρασμα ήταν ότι είμαστε ενωμένοι μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις. Είχαμε και δύο συνεδριάσεις, ε, αυτό που αποκαλούμε πίεση ε, ναι, είναι οι εταίροι έτοιμοι για προσχώρηση, αλλά επίσης ε, τα μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, έντονα βρισκόμαστε πίσω από την, υποστηρίζουμε απόλυτα την ΟΣΥΗ και την προσπάθεια αποστολής, ε, αποστολών, ανάπτυξη αποστολών από πλευρά τους, τους ε, εξασφαλίζουμε τα οχήματα προστασίας, ε, χρηματοδοτούμε επίσης τις δράσεις τους και χθε ε, βλέπαμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να υποστηρίξουμε τι εναλλακτικέ δυνατότητε. Τρίτον, ξεκινήσαμε τώρα την αποστολή μα ώστε να βοηθήσουμε <clears throat> την μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλεια, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική ασφάλεια σε σχέση και με την Ουκρανία. Και τέταρτον, υπάρχει το θέμα <clears throat> το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί μια και δεν έχουμε ακόμα συμφωνία και δεν υπάρχει βούληση με τα όπλα να δράσουμε. Φυσικά το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι κυρώσει ει βάρος της Ρωσίας. Δύο παρατηρήσεις γι' αυτό. Πρώτον, φαίνεται ότι έχουν επιπτώσεις και επηρεάζουν την κατάσταση οι κυρώσει. Και στο Ιράν νομίζω, χάρη στις κυρώσεις μπορέσαμε να προχωρήσουμε με τους Ιρανούς και έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις που προχώρησαν με αυτούς. Αλλά επίσης και αυτό το οποίο είναι το οποίο εκπλήσει είναι το ότι παρόλες τις κυρώσεις και παρόλο το πλαίσιο των κυρώσεων, οι κυρώσεις πλήττουν και εμάς, έχουν επιπτώσει σε εμάς. Και για την διασφάλιση εσωτερικής ε, ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, αν λέγατε πριν από κάποια χρόνια ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει τέτοιες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, θα έλεγε κανείς είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, απίθανο. Και όμως έγινε. Τώρα, Έχουμε φυσικά και το θέμα της ε, αναχέτησης του ΙΚΙΣ, ε, του Ισλαμικού κράτους Ιράκ και Συρίας ε, και με βάση το συνασπισμό της Συμμαχία υπό την ηγεσία των ΙΠΑ. Καλό είναι ότι οι χώρες στην περιοχή, τα Εμμυράτα για παράδειγμα και άλλοι συμμετέχουν όπως και η Σαουδική Αραβία, ένα διαφορετικό, απόλυτα διαφορετικό σκηνικό από τον πόλεμο που είχαμε στη Λιβύη ή και παλαιότερα στο Ιράκ. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπου οι αλλοδαποί μαχητές που βρίσκονται πολύ ψηλά στην ημερησία διάταξη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων ασχολήθηκαν, υιοθετήθηκε μόλι μια στρατηγική καταπολέμηση τη τρομοκρατία και με του συναδέλφου Κόζη για την εσωτερική ασφάλεια θα έχουμε ε, συνάντηση μαζί του να δούμε πώ θα μπορέσουμε κατά τα μέσα Νοεμβρίου να δούμε η στρατηγική αυτή πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Έχουμε και το θέμα, για παράδειγμα, του τι γίνεται και με τα θέματα των, ε, ε, ε, της λαθρεμπορίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορεί να παρασχεθεί όσον αφορά την Συρία. Πολλοί πρόσφυγες βρίσκονται από τη Συρία στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία και σε άλλες χώρες και υποστηρίζουμε την περίθαψη αυτών των προσφύγων με κονδύλια Υπάρχει και το θέμα της στρατιωτικής δράσης ε, που μπορεί ίσως να είναι αναγκαία αλλά δεν είναι η μόνη λύση. Πρέπει να υπάρχει και πολιτική λύση. Στο Ιράκ για παράδειγμα είναι σαφές ότι πολλά από αυτά τα οποία συνέβησαν με το Ίκης είναι επίσης το αποτέλεσμα έλλειψης ενδιαφέροντος από πλευράς της κυβέρνησης Αλμαλίκη όσον αφορά την σουνητική μειονότητα σε κάποιες περιοχές της χώρας στο Ιράκ. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά και να βοηθήσουμε τις χώρες που είναι όμορες χώρες και έχουν σύνορα προς τη Συρία, Ιορδανία, Λίβανο, καταπολέμηση τρομοκρατίας. Ε, παροχή ε, ανθρωπιστικής ε, βοήθειας αλλά επίσης και υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου μέσω μιας ξεχωριστής δράσης που θα, δεν θα προβλέπεται από την ΚΕΠΑ αλλά θα χρηματοδοτείται από τα κονδύλια της Επιτροπής για τη λωρίδα της Γάζας φυσικά και είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός λοιπόν και να υποστηρίξουμε μια ολοκληρωμένη συνολική προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την επίλυση προβλήματο του προβλήματος με τις αποστολές που έχουμε εκεί επιτόπου και την εκπροσώπησή μας επιτόπου. Έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις στο τραπέζι. Η Λιβύη παραμένει μια τεράστια πρόκληση πολλές σειράξεις ε, και συγκρούσεις μεταξύ Ισλαμικών δυνάμεων και άλλων δυνάμεων υπήρξαν ε, στην Λιβύη. Έχουμε και την αποστολή μας ε, στην Λιβύη που έπρεπε να μειώσουμε όσον αφορά τα στελέχη και μετατέθηκαν στην Τινησία διότι υπήρχαν προβλήματα ασφάλειας και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον όταν όλοι συγκρούνται με όλους όπως συμβαίνει στη Λιβύη και πρέπει να δούμε και τους γείτονες των γειτόνων μας, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για παράδειγμα, όπου έχουμε και την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, μια γερφυροποίηση όσον αφορά την δράση των Ηνωμένων Εθνών και έχουμε τρεις μήνες που θα καταστεί δυνατή αυτή η γεφυροποίηση, η μεταβατική περίοδος. Να δούμε επίση πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη μέσα στον τομέα, στο πλαίσιο του τομέα ασφάλεια, όπου έχουμε διαφορετικέ εναλλακτικέ λύσει που εξετάζουμε και πρέπει να εξετάζονται. Και πρέπει να υπάρξει και ένα καλό συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το πεδίο. Επίση, η ιδιαίτερη εμπλοκή στην υποσαχάρια Αφρική, στη ζώνη της Σαχέλ και με μια αποστολή για την υποσαχάρια Αφρική και το Μαλί για να βοηθήσουμε τις πολιτικές και δυνάμεις ασφαλείας. Φυσικά η αποστολή μας έχει το ίδιο περίπου εύρος όπως και στον Νίγηρα. Και εκεί πρέπει να δούμε το ίδιο, τα ίδια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε, τρία θέματα. Το κέντρο επιχειρήσεων, OP Center. Ίσως τα έχετε δει αυτά για το μέλλον αυτού. Έχουμε λάβει πολιτική απόφαση στην πίεση να παραταθεί η εντολή ώστε να ευθυγραμμιστούμε με την εντολή των ε, ε, αποστολών που παρακολουθούμε στενά. Έχει επεκταθεί η εντολή μέχρι το 2016 τώρα, αλλά και γεωγραφικά έχει επεκταθεί στο σύνολο της Αφρικής συγγνώμη, στην υποσαχάρια ζώνη της Αφρικής διότι αυτό θεώρησαν τα κράτη-μέλη ότι αυτό θα οδηγούσε σε πρόσθετη αξία, δημιουργία πρόσθετης αξίας και ωφέλους ε, Είχα αναφέρει ήδη στην αρχή ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να αναπτύξουν το δικό τους δυναμικό ξεχωριστά, κάτι που κάνουμε σε σχέση με την Αφρικανική Ένωση, με αυτό που κάνουμε με την αρχιτεκτονική για την ειρήνη στην Αφρική και την αρχιτεκτονική της ειρήνευσης. Φυσικά όμως και με τις δυνατότητες που παρέχονται για κονδύλια όσον αφορά για παράδειγμα το Μάλι που γίνεται καλή δουλειά για να αναχαιτήσουμε και καταπολεμήσουμε την Σαμπά. και επίσης ε, και μια συνάντηση με Αφρικανούς εταίρους και Αφρικανούς ε, συναδέλφους ε, που είναι καλό νομίζω και μια κοινή αποστολή στο Μαλί που έχουμε αποστολή εκεί και τα Ηνωμένα Έθνη που είναι παρόντα εκεί είναι σημαντικό να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις ε, και βιώματα μεταξύ μας. Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό η κατάρτιση, η ανάπτυξη δυναμικού και δυνατοτήτων από πλευρά των εταίρων ώστε να είναι σε θέση εκείνοι να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τα θέματα ασφάλειας από πλευρά του. Και είναι σαφές ότι πρέπει και το θέμα του εξοπλισμού να εξεταστεί και να καλυφθεί. Υπάρχει τώρα μια πρωτοβουλία Train and Equip ε, κατάρτισης και εξοπλισμού. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι δυνατόν με κοινοτικά μέσα και μέτρα να γίνει αυτό. Αποκλείεται από τις συνθήκες της Αβώνας. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους και διόδους για να το κάνουμε. Ίσως μακρηγόρησα φοβούμε, αλλά προσπάθησα να, με αδρές γραμμές να σκιαγραφίσω το τι συμβαίνει. Συνεχίζεται το έργο, βρίσκεται υπό εξέλιξη. Work in progress, έργο υπό εξέλιξη. Αλλά πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, προχωρήσουμε. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πεσβευτά για αυτή την πλήρη εισαγωγή που κάνατε. Θα σας τεθούν πολλές ερωτήσεις πιστεύω. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στους συντονιστές, επιτρέψτε μου να θέσω τη δική μου ερώτηση. Άκρος ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Ακούσαμε τον, τα όσα μας είπε για την άποψη του πίεση. Αναφερθήκατε σε νέες απειλές, σε παλιές μακροχρόνιες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εγώ προσωπικά σας είμαι ευγνώμων για την παρουσίασή σας, για την παρουσίαση της καταστάσεως στην ε, Αφρική που είναι και το επίκεντρο των συζητήσεών μας στις συνεδριάσεις μας της Υποπιτροπής οι τελευταίοι μήνες έχουν αφιερωθεί στη συζήτηση των απειλών που δημιουργεί το ISIL, το ΙΚΙΣ στα ελληνικά διότι επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν το χαλιφάτο. Λίγο πολύ είμαστε ενωμένοι στην προσέγγιση για τις απειλές που τίθει, τίθονται από το ISIS ή οίκη στα ελληνικά. Θα ήθελα να ακούσω την παρουσίασή σας όσον αφορά την πολιτική προσέγγιση, διαμόρφωση πολιτικής για δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι αυτής της απειλής πολιτική που αφορά ε, εσωτερικές απειλές που δημιουργούνται από πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως που μάχονται εντός των τάξεων του ISIS. καθώς και ποιες είναι οι γεωπολιτικές προκλήσεις που δημιουργούνται. Χθες μπορέσαμε να, ακούσαμε την, ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Μπαρζάνη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας για την κατάσταση στην περιοχή. Όμως είχαμε και διαφορετικής απόψης όταν συζητήσαμε το ΕΝΚΕΠΑ και τις ευρωπαϊκές δυνατότητες που υπάρχουν και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων υπάρχει μια νέα κατάσταση που διαμορφώνεται ανατολικά μετά την ανοιχτή επιθετικότητα της Ρωσίας που εκδηλώθηκε στην Ουκρανία και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η απόψή σας επ' αυτού. Έχουμε από τη μία πλευρά πολύ σκληρή ρητορική που χρησιμοποιείται, αποφάσεις, δηλώσεις κλπ. Λαμβάνονται αποφάσεις οικονομικής φύσεως για οικονομικές κυρώσεις για την ώρα. Ε, όμως για, συνεχίζουμε όμως ανοιχτά να συνεχίζονται διάφορα διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με τους, ε, αυτούς τους εχθρικούς μας γείτονες. Σε λίγο συζητήσουμε το Γαλιλαίος και υπάρχει και σαφής συνεργασία με τη Ρωσία εκεί και υπάρχουν και άλλες σχέσεις και για τις ομάδες μάχης υπάρχουν κάποιες πτυχές συνεργασίας με τη Ρωσία ε, για τα battle groups ποια είναι η πολιτική προσέγγιση όσον αφορά αυτού του είδους τις προκλήσεις. Αυτό ήθελα να θέσω. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Να δώσω το λόγο τώρα στους συντονιστές. Ο κύριος Γκάλερ, εκ μέρους του ΕΛΚ, πρώτα απ' όλα, έχει το λόγο. Yeah. Um, Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη Στίβενς για το ευρύ φάσμα αυτής της παρουσίασης που βρισκόμαστε σήμερα. Ίσως μια εκπροημίου παρατήρηση. Αν πραγματισμός, ρεαλισμός σημαίνει ότι θα αντιδρούμε επαρκώς στο σωστό μέτρο στις κατεπίγουσες καταστάσεις, τότε μπορώ να δεχθώ αυτή την προσέγγιση του πραγματισμού, να έχουμε μια σωστή αντίδραση. Αν όμως πραγματισμός σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να παρελκύσουμε ώστε να μην υπάρχει υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών και στόχων, τότε δεν θα συμφωνούσα με μια τέτοια προσέγγιση. Αυτός ε, παρατήρησε εκ προημίου. Η εντύπωσή μου είναι από τα όσα ε, αναφέρθηκαν, ότι σαφώς ένα υψηλότερο επίπεδο έχετε φιλοδοξίας από ότι η προκατοχό σας και για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αυτό με σαφή τρόπο αναφέρθηκε να παίξετε σκληρό παιχνίδι αναφέρθηκε όπως είχε πει. Και ελπίζω λοιπόν ότι με αυτή την προσέγγιση η συνένεση των κρατών μελών θα μπορέσει πιο έντονα να ενισχυθεί ώστε η πατή εκπρόσωπος να μπορεί άμεσα δραστήρια να προσπαθεί να παρακολουθεί τα πράγματα και όχι να δει αν κάτι τυχαία απορρέει. Θα ευχόμουν λοιπόν η απέτηση αυτή, η διεκδίκηση αυτή να γίνει πραγματικότητα. Για τις ερωτήσεις που έχω. Καταρχήν κάτι πιο συγκεκριμένο να αναφερθεί για τη συζήτηση για το μηχανισμό Αθηνών. Πού βρισκόμαστε σχετικά. Είπατε ότι βρίσκονται προτάσεις στο τραπέζι επιτραπέζης. Ίσως μπορούν να ε, αποσαφινιστούν αυτές, να δούμε τι συμβαίνει. Διότι στην ίδια την πραγματικότητα τι διαπιστώνουμε. Κάποια κράτη-μέλη για αυτό το λόγο δεν συμμετέχουν σε σχέση με τη διάθεση ενόπλων δυνάμεων επειδή δεν είναι ε, ικανοί να, ικανά να πληρώσουν 100% όμως το ευρωπαϊκό ποσοστό μπορούν να το συγχρηματοδοτήσουν από πλευρά του και έτσι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σωστά. Ε, απαιτείται λοιπόν να καταλήξουμε σε μια τέτοια κατάσταση ώστε στο τέλος τέλος σε σχέση με τις διατάξεις ε, του μηχανισμού αυτού το υλικό, τον εξοπλισμό σε πρώτη φάση αλλά και τι ένοπλες δυνάμεις, το έμψυχο υλικό να μπορούμε να διαθέσουμε σε μια κοινή χρηματοδοτούμενη, κοινά χρηματοδοτούμενη δράση μέσα από ένα κοινό ταμείο αυτό θα το θεωρούσα σημαντικό, διότι ακριβώς τα μεγαλύτερη κράτη που θεωρητικά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, τέτοιο όλο και πιο συχνά θα δρούσαν. Τα μικρότερα θα είχαν διαθέσιμους στρατιώτες αλλά δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν δράσεις. Θέλω να γνωρίζω τι επακριβώς βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως δυνατότητα. Και τώρα για την διαφρομένη συνεργασία πράγματι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν δείχνει ότι σε συγκεκριμένα πράγματα μπορεί κανείς να προχωρήσει παρακάτω. Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το μέσο. Θα ήταν λοιπόν, άξιζε τον κόπο να εντείνουμε τη συζήτηση και να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πούμε ορίστε εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα operation ή headquarters ή κάτι άλλο όπου κάποια κράτη-μέλη ή όπου όλα σχεδόν λένε να προχωρήσουμε αλλά εντάξει θα πρέπει να πει και η Μεγάλη Βρετανία εντάξει ε, δεχόμαστε ότι θα προχωρήσετε εσείς αλλά εμείς δεν θα συνεχίσουμε διότι μπορεί έτσι να παραμείνει λοιπόν να υπάρξει αυτή η διαφωνία αλλά οι άλλοι να συνεχίσουν επ' αυτού. Το άλλο θέμα τώρα, στην ενδιάμεση περίοδο μεταξύ των δύο κορυφών, Δεκέμβριο 2013 και Ιουνίου 2015, πού βρισκόμαστε ακριβώς σε σχέση με την υλοποίηση του έργου μας, των καθηκόντων που έχουμε αναλάβει και επομισθεί. Μπορούμε δεδομένων των αλλαγών στην παγκόσμια κατάσταση στο παγκόσμιο τοπίο στην γειτονία μας να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με πιο φιλόδοξο τρόπο θα θελήσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία αποφασίζονται. Αυτό θα ελπίζα να μπορούσε να γίνει διότι αντί για ένα δακτύλιο φύλων, μια αλυσίδα φύλων ή ένα δακτύλιο συμμάχων, έχουμε ένα δακτύλιο πυρός, δακτύλιο φωτιάς γύρω μας και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Are other members willing to, to ask Λοιπόν, άλλος που θέλει να θέσει ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Πρέσβη, αν θέλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση και μετά συνεχίζουμε σε άλλο γύρο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Είναι πολύ ε, σχετικές με τη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω με την τελευταία. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την εφαρμογή των καθηκόντων που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013. Αναφέρθηκα λίγο σε αυτό το θέμα στην εισαγωγή μου ότι πράγματι ε, όσον αφορά την ορατότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεών μας είχαν θεθεί κάποιοι στόχοι και το δυναμικό και τη βιομηχανική βάση. Έχουμε και την έκθεση τη κάθε άστον του Σεπτεμβρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Αλλά πρέπει να πω ότι περνάμε πολύ σημαντικές στιγμές, ε, είναι σημείο καμπή, τώρα, αλλά πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά ακόμα. Και το, σαν πρόεδρος του SPC είδα ότι δεν είναι πάντα εύκολη η συζήτηση. Αν θέλει κανείς να βελτιώσει τη χρηματοδότηση των αποστολών και των επιχειρήσεων, τα κράτη-μέλη έχουν διάφορες απόψεις. Αν μιλήσουμε για τις μάχημες μονάδες, συγκροτήματα μάχης που ήταν στοιχείο της ταχείας δράσης, αυτό πάντα συζητείται σαν θέματα, συναντώνται οι διάφοροι υπουργοί και οι πολιτικοί διευθυντές ε, στο PSE. Ε, πολλή κουβέντα αλλά λίγη πρόοδος. Ε, πολλά από μένα γίνουν. Όπως ανέφερα, υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου έχει σημειωθεί πρόοδος, όπως η στατική τη θαλάσσια ασφάλεια, σημαντική δουλειά έχει γίνει. τώρα προσπαθούμε να ετοιμάσουμε ανάλογο σχέδιο δράσης. Θα συζητηθεί στο PSC e τις επόμενες εβδομάδες για την κυβερνοασφάλεια το ίδιο. Πολλά έχουν γίνει και εκεί εκπαίδευση και ο εξοπλισμός, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όσον αφορά τον εξοπλισμό και εκεί έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδο. Δεν είναι εύκολο όμω να βρεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι. Θα συζητηθεί και αυτό στο PC. Η γενική τάση ποια είναι. Ότι είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Ακόμα και στα βασικά ανεφοδιασμός, σε βασικές προσπάθειες ανεφοδιασμός, όπου ηγούνται κάποιες χώρες, η Ολλανδία και η Ιταλία, παραδείγματο χάρη, η Γαλλία, στο θέμα αυτού. Υπάρχει κάποια πρόοδος, όμως ε, γίνεται σταδιακή πρόοδος, βήμα-βήμα. Ε, πράγματι ε, υπάρχει πολλή δουλειά που απομένει να γίνει και νομίζω ότι οι Υπουργοί το Νοέμβριο θα δώσουν μεγαλύτερη ορμή στην προσπάθεια. Τι βλέπω πάντα, ότι στο επίπεδο των ηγετών, των υπουργών, και το έχω προαναφέρει και αυτό σε άλλες συναντήσεις, Θέλουν να υπάρξει κοινή χρήση των μέσων. Το pooling and sharing θέλουν να το προωθήσουν. Ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε και να συνενώνουμε το δυναμικό κάθε χώρας γιατί μειώνεται παντού το δυναμικό. Όσον αφορά όμως ε, την, στους ειδικού για τα θέματα άμυνας τα περιπλέκεται η κατάσταση. Δεν λέω ότι δεν επιτυγχάνεται πρόοδος αλλά είναι επώδυνη, δύσκολη. Όσον αφορά το δεντρολογικό κώδικα ε, και εκεί υπάρχει συμφωνία μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών για τον, και τη CDA για τον διοντολογικό κώδικα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ε, πού βρισκόμαστε. Ε, νομίζω ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Ελπίζω ότι είναι μισογεμάτο. Υπάρχει δουλειά ακόμα πρέπει να γίνει, τόσο ώστε και το υπόλοιπο ποτήρι να γεμίσει. Όσον αφορά το ΠΕΣΚΟ, ε, δεν είναι θέμα που αφορά διαμάχη μεταξύ κρατών μελών. Ε, δεν είναι επιτραπέζης αυτό. Κανείς δεν συζητά τι γίνεται με το θέμα αυτό για το ΠΕΣΚΟ. Είναι ένα από τα νέα στοιχεία της συνθήκης που ίσως θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον αφορά και το ότι δεν θα κινηθούμε όλοι μαζί, ίσως να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, κάποιες ομάδες χωρών ε, να προχωρήσουν ε, μόνες τους πρώτες. Υπάρχει όμως, έχετε δίκιο, παρακαλώ να αποφεύγετε το διάλογο λέει η Πρόεδρος, δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κινούμεθα μαζί, Κάποιοι μπορούν να προχωρήσουν ταχύτερα και να ζητήσουν από άλλους να ενωθούν μαζί τους. Όταν είχε γίνει πρόταση, είχε γίνει μια συζήτηση και υπήρχε διαφοροποίηση των Υπουργών, υπήρχαν πολλές απόψεις. Έκτοτε δεν ακούω κάποιον να το προωθεί το θέμα, παρόλο που πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα de facto, υπάρχει συνεργασία το PESCO de facto. Ε, ε, ίσως να υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν ε, ιδεολογικές διαφορές κρατών μελών. Όσον αφορά το Αθήνα, δεν είμαι 100% δεν έχω γνώση, πλήρη γνώση των λεπτομεριών. Από ό,τι κατάλαβα δεν απέχουμε πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα και συνδέεται η δυσκολία με το κοινό κόστος και τι μπορούμε να εντάξουμε στο κοινό κόστος εάν ε, στέλνει κανείς μια, έχει καμία στρατιωτική επιχείρηση, ε, δύσκολος ο προσδιορισμός του, του κόστους. Όλοι ζητούν από εμά να υπομισθούμε το κόστος. Η, η, Γαλλία κάνει πολλά, στο Μαλί και λοιπά δεν υπάρχει ο επιμερισμός και αλλού κινούνται άλλες χώρες και υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μπορούμε να τα βάλουμε στο κοινό κόστος. Θέλουμε να αυξήσουμε τις κοινέ δαπάνες ούτω ώστε το οικονομικό βάρος των προσπαθειών να μοιράζεται σε μεγαλύτερο αριθμό μελών, κρατών μελών. Και βέβαια έχουμε εκείνους που συμβάλλουν περισσότερο και τα κράτη-μέλη εκείνα που λένε ότι ε, ε, ε εμείς έχουμε τα περισσότερα στατεύματα ε, που διαθέτουμε επιτόπου, αναπτύσσουμε επιτόπου και δεν θέλουμε να πληρώνουμε δύο φορές και μετά να συμβάλλουμε οικονομικά στο μηχανισμό Αθήνα ε, και, για να αυξηθεί το κοινό κόστος. Ε, είναι παράδοξη κατάσταση. Και εκεί ε, πρέπει να γίνει κάποια δουλειά και βέβαια είμαστε στο, στη δεύτερη περίοδο που θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, για την πολιτική προσέγγιση, το ερώτημα της Προέδρου, όπως σας είπα, η κοινή πολιτική άμυνας και ασφαλείας χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση βέβαια όσον αφορά το ISIL υπάρχει ε, κοινή συνιστόσα πρώτα απ' όλα χρειάζεται μια άμεση κατεπίγουσα ε, ανάγκη να συγκρατήσουμε την, ε, ε, την ISIL με τους βομβαρδισμούς που γίνεται με τη συνεργασία με έξι χώρες και με συνεργασία με τις χώρες της περιοχής πολύ σημαντικό όμως είναι να δούμε και το πολιτικό μέτωπο ε, στο Ιράκ. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε αυτή η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση ε, να μπορέσει να ε, συμπεριλάβει πολλές συνιστώσεις και οι Σουνίτες και οι Κούρδοι να αισθάνονται ότι μπορούν να συμμετάσχουν άνετα. Κάτι που δεν ίσχυε παλιά, όπως σας είπα, παλιά η κυβέρνηση του Αλμαλίκη αγνοούσε κάποιους, κάποιες περιοχές του Ιράκ, σουνιτικές περιοχές του Σουνίτες αμέλησαν. Ε, τους είχαν ε, πράγματι αμελήσει. Σχεδόν τους οδήγησαν στη φτώχεια. Δεν είχαν καμία άλλη εναλλακτική παρά να πολεμήσουν. Και Άισιλ βρήκε ε, έφορο έδαφος εκεί και προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από το Άισιλ γιατί πραγματοποιούν μαζικές δολοφονίες και εκτελέσεις και κάποιες φυλές πολεμούν τα Άισιλ. και αναφερθήκατε στους ξένους μαχητές που είναι βασικό πρόβλημα στο θέμα αυτό και για τους Υπουργούς Εξωτερικών και τους Υπουργούς Εσωτερικών, διότι έχουμε εκείνους που φεύγουν και ενισχύουν τις δυνάμεις του Άσυλ και είναι αξιοσημείο το φαινόμενο, διότι ε, όταν ε, σχετίζεται και με το Ισλάμ αλλά και με άλλα στοιχεία έχω την εντύπωση το φαινόμενο βλέποντας τις εικόνες εκείνων που αποκεφαλίζονται ε, δεν φαίνεται να τρομάζει εκείνους που κινούνται προς την περιοχή. Ε, το συζητούσαμε με τον Τούρκο πρέσβη που διαπιστώνει ότι υπάρχει το ίδιο φαινόμενο. Σχετίζεται ε, με ανθρώπους που τους δίνουν ένα όπλο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και τους δίνει κανείς ένα όπλο και τους στέλνει στη μάχη και ξαφνικά ανήκουν σε κάποια οργάνωση που προδεύει και αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ ισχυρό. Ε, και αυτό είναι κάτι που προσελκύει κάποιους από αυτούς που πάνε και στρατολογούνται. Και βέβαια, βέβαια θα επιστρέψουν και όλες οι χώρες, το Υπουργείο Εσωτερικό και Δικαιοσύνη το συζητούν αυτό το πρόβλημα. Τι γίνεται όταν επιστρέψουν και έχουν στρατηγική αντιτρομοκρατία στο εσωτερικό μέτωπο, αντιτρομοκρατική πολιτική και στις εξωτερικές ε, σχέσεις θα πρέπει οι εξωτερικές σχέσεις να δημιουργήσουν συμπράξεις με διάφορες χώρες όπως η Τουρκία που είναι χώρα κλειδί και η Τουρκία πρόσφατα έχει κάνει πολλά πράγματα. Δεν ήταν τόσο δραστήρια σε κάποια φάση στην αρχή η Τουρκία αλλά τώρα νομίζω ότι καταβάλει πολλές προσπάθειες θα πρέπει να συμμετάσχει ούτως ώστε να μην υπάρχει μετακίνηση ανθρώπων να μην πηγαίνουν στο ISIL αλλά να δούμε και τι γίνεται με εκείνους τους μαχητές του ISIL επιστρέφουν στην, επιστρέφουν Ευρώπη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό μέτωπο. Χώρες μου όπως η χώρα μου το Βέλγιο λαμβάνουν μέτρα ούτω ώστε να συνεπάγεται κάποιο κόστο όταν κάποιος πηγαίνει να πολεμήσει με, στο Άσυλ, να φερείται το διαβατήριο, κάποια επιδόματα κλπ. Ε, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των δικών μας υπηρεσιών, των υπηρεσιών ασφαλείας, εσωτερικής ασφαλείας και των τουρκικών υπηρεσιών να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση, να παρακολουθούν του κατάλληλου ανθρώπου. Συνεχίζονται οι προσπάθειε στο εξωτερικό μέτωπο. Πρέπει να δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσει και με την Τουρκία αλλά και με άλλε χώρε. Βέβαια υπάρχει και το άλλο θέμα. κάποιοι στι χώρε τη περιοχή επίση οικονομικά έχουν στηρίξει κάποιες από αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να δούμε ε, τι μπορούν να κάνουν οι χώρες σχετικά με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό χώρες Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, το Κατάρ κλπ ε, που να ανήκουν στη συμμαχία που πολεμά το ISIL. Καμιά φορά όμως η εικόνα είναι κάπως ανάμεικτη όσον αφορά αυτό το θέμα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Τεράστιο θέμα, ανθρωπιστικό βάρος, τεράστιο ανθρωπιστικό βάρος στη Συρία ο αριθμό των εκτοπιστέντων, εσωτερικά εκτοπιστέντων ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλος και καθημερινά βλέπουμε τα δεινά που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι και βέβαια έχουμε Λίβανο, Ιορδανία και σε αυτές τις χώρες, στο Λίβανο έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Ε, έχουν κλείσει τα σύνορά τους δυστυχώς για τους πρόσφυγες στο Λίβανο δεν μπορούν να τα καταφέρουν να ανταποκριθούν πλέον. 1,5 εκατομμύριο στην Τουρκία, μισή από αυτού είναι σε στατόπεδα, 500.000 περίπου είναι στα στατόπεδα, οι υπόλοιποι είναι στην κοινωνία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 600-700.000 άνθρωποι να μπαίνουν στην κοινωνία σα, νερό, σχολεία, ε, υγεία κλπ. Καταλαβαίνετε. Ανταγωνισμό στην αγορά εργασία, άρα έχει αντίκτυπο για τι χώρε, για την Ορδανία, η οποία ήδη είναι αρκετά προβληματική σαν χώρα. Η Ορδανία ο Λίβανος και η Τουρκία έχει προβλήματα παρόλο που η Τουρκία είναι πολύ αρκετά δύσκολος εταίρος και η προσέγγιση μας όσον αφορά τη Ρωσία. Α, συζητήθηκε εκτενώς αυτό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τη Ρωσία ε, είναι να ακολουθήσουμε διτή προσέγγιση. Δηλαδή από τη μία πλευρά να αυξήσουμε το κόστος για την πολύ κακή συμπεριφορά των εισαγωγικών της Ρωσίας που παραβίασε κάθε κανόνα επιβάλλοντας κυρώσεις όπως είπα δεν νομίζει ότι ήθελε κανείς να χρησιμοποιήσει όπλα, αυτό είναι σαφές. Η Ρωσία όμως χρησιμοποιεί καμιά φορά ισχύ, αλλά ο μηχανισμός των κυρώσεων έχει προχωρήσει αρκετά, έχουν προχωρήσει αρκετά μακριά, είναι κυρώσεις που πλήττουν και τις δικές μας χώρες. Εγώ ε, υπάρχουν, ε, αν πάτε στην Ήπεθρο θα δείτε ότι υπήρχαν κάποιοι γεωργοί που εξήχαγαν στη Ρωσία πρέπει να βρουν άλλη εξαγωγική ε, αγορά. Πληττόμεθα κι εμείς. Αυτό που μας εκπλήσει είναι ότι στη νέα κατάσταση ίσως χάρη σε αυτή τη νέα κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ενωμένη σαν ένα μπλοκ, μια ομάδα ακόμα και με δύσκολες κυρώσεις. Χώρες όπως η Ιταλία, η Κύπρος έχουν ε, πολλά συμφέροντα στη Ρωσία. Η οικονομία τους ε, έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία και έλαβαν και αυτές εφάρμοσαν κυρώσεις. Τώρα ε, έγιναν οι εκλογές όπως αποκαλούνται οι εκλογές στο, στο, στις δύο το Λουγκάνσκ που θεωρούνται παράνομες και δεν αναγνωρίζονται και σίγουρα ε, ίσως να είναι εμπόδιο για την ειρήνη και είχαμε και συζητήσει στο PSC e και δημιουργήθηκε εντύπωση ότι πρέπει να δούμε μήπως πρέπει να προσθεθούν και άλλα ονόματα στον κατάλογο εκείνων στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να κλείσουμε τις πόρτες. Θα πρέπει να συνεχιστούν ε, συνομιλίες με τη Ρωσία, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε είναι επικίνδυνη ή όχι. Είναι μια μεγάλη χώρα, ε, είναι μια υπερδύναμη, πολύ ισχυρή χώρα δίπλα μας. Και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά να συνομιλούμε μαζί τους και εκείνοι βέβαια ε, έχουν άλλη αντίληψη για την ισχύ. Χρησιμοποιούν κάθε είδους ε, τέχνασμα και τεχνική που εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για την ώρα. Ίσως ε, δεν ξέρω αν αρκεί η απάντηση αυτή στην ερώτησή σας. Είναι εντελώς νέα κατάσταση. Μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πετύχει κάτι καλό για την Ουκρανία και πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ δύσκολο ο δρόμο τη μεταρρύθμιση και πολύ δύσκολη η περίοδος που περνά η χώρα, αλλά προσπαθούμε με τη Συμφωνία σύνδεση να βοηθήσουμε και με την πλήρη αυτή εμπορική συμφωνία, όμω από την άλλη πλευρά γίνεται αυτό αντιληπτό σαν ε, ε, σαν, ε, μάλλον είναι σαν να, πατήσαμε, τη μεγάλη αρκούδα και η αρκούδα οργίστηκε. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, ε, υπάρχει μια διαπάλη, μια διαπάλη κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και ο κύριος Γκάλερ και εγώ θα μπούμε σε λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά, αλλά επιτρέψτε μου καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Στέτινα που θέλει να θέσει κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για την Ουκρανία πιο συγκεκριμένα. Οι σειράξει μεταξύ ε, ρωσικών, φιλορωσικών και αντιρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντανιέτσκ δείχνουν ένα πράγμα. Αφενός ε, έχουμε την εμπλοκή των ε, Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και αφετέρου τις εθελοντικές δυνάμεις μεραρχίες εθελοντών. Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σήμερα δεν είναι ελεύθερης βούλησης ε, αυτές οι δυνάμεις. Ε, βρίσκεται σε ικτρή κατάσταση ο Ουκρανικός στρατός. Έχουμε μετακομμουνιστικούς στρατηγού ε, που είναι στα ενία στην Ουκρανία ακόμα και η διαφθορά είναι υψηλού επίπεδου. Νεότατοι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί και καταρτιστεί παίρνουν όπλα και συμμετέχουν στις σειράξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυχώς συμμετέχει στην καταπολέμηση τρομοκρατίας στην Αφρική. Διαρωτώ με, γιατί δεν έχει την ίδια επιτυχία η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Αυτή είναι η συγκεκριμένη μου ερώτηση για αυτό το θέμα. Πώς δεν βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ουκρανούς στην Ουκρανία μέσω συγκεκριμένων παροχών οπλισμού, εξοπλισμού όπλων ώστε να δράσει η Ουκρανία αποτελεσματικά έχει είναι βεβαρημένη η κατάσταση. Με απλά καλάσνικοφ, με απλά αυτόματα όπλα πολεμούν οι Ουκρανοί κατά των Ρώσων και δεν μπορούν με τα καλάσνικοφ να κερδίσουν τη μάχη. Φυσικά δεν πρέπει εμείς οι ίδιοι να συμμετάσχουμε με δικές μας ένοπλες δυνάμεις, αλλά μπορούμε με εξοπλισμό και όπλα να υποστηρίξουμε τον αγώνα των Ουκρανών. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Επανέρχομαι. Πιστεύω τον Μπάστ ε, δεν πήγα εκεί θέλοντας να συμμετάσχω. Ήθελα να διατηρηθεί ο διάλογος να επικρατήσει ειρήνη και αν αρνηθούμε κάθε ύπαρξη συνομιλητού ε, για να συνομιλήσουμε δεν υπάρχει δυνατότητα να καθίσουν τραπέζι διαπραγματεύσεων οπότε είναι πόλεμος μέχρι τέλους αλλά θα πρέπει να επιστρέψει η ειρήνη το ερώτημά μου δεν αφορά αυτό το θέμα όμως είδα αυτή τη, τη, τα σχολεία που βομβαρδίστηκαν εκατοντάδες σχολεία μου είπαν ότι βομβαρδίστηκαν μπορώ να πω ότι είδα είδα νοσοκομεία βομβαρδισμένα όπου επέλεξαν συγκεκριμένα, δεν θέλω να ξέρω ποιος, δεν θέλω να, να πω ποιος είναι υπεύθυνο, αλλά επέλεξαν, δεν θα τοποθετηθώ. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι ο πληθυσμός είχε τρομοκρατηθεί, ε, ε, διαπίστωσα πέρα εκτός αποστολής ε, πήγα και μίλησα με τον κόσμο και κατά την άποψή μου θέλουν να διατηρηθεί η ακαιρεότητα, η εδαφική κυριότητα της Ουκρανίας. Αυτό δεν το συζητούν, το αφισβητούν. Αλλά διαπιστώνω ότι αυτό που μου είπε ο καθένας και γυρίζαμε ταινία εκείνη την ώρα. Όλοι μου είπαν ότι δεν είναι πλέον δυνατόν. Πώς να αποφευθεί η τρομοκρατία με κάποιο τρόπο και δεύτερο, πώς να, να υπάρχουν σχέσεις, να διατηρηθούν οι σχέσεις και να διατηρηθεί η, χώρα και να κινηθεί προς την ειρήνη. Τι μπορούμε να κάνουμε. Εν αυτή τη ενία λέω ότι η μία αναγνώριση των εκλογών δεν είναι πολύ συνετό. Θα πρέπει να βρούμε άτομα στα ανατολικά της Ουκρανίας με τους οποίους να υπάρξει συζήτηση θα πρέπει να αναγνωριστεί μια νομιμότητα. Από την αρχή λέμε ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν καμία νομιμότητα, είναι τρομοκράτε. Τι θέλετε να κάνουμε. Δεν μπορούμε πλέον να έχουμε διάλογο ειρηνευτικό. Πώ θα βρείτε λύσει, πώ θα βρούμε λύσει για να πάμε προ την ειρήνη. Αυτό είναι το θέμα. Η κυρία Αναγκόμες. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω από την αρχή γιατί έπρεπε να είμαι σε μια άλλη επιτροπή και δεν μπόρεσα να ακούσω την αρχή των παρεμβάσεων. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ κάθετα με αυτά που μόλις ελέγχθησαν. Δηλαδή το να αναγνωρίσει κανείς αυτές τις ε, πλαστές, τις νοθευμένες εκλογές στην Ουκρανία. Βεβαίως και πρέπει να διατηρηθεί ο διάλογος, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτι το οποίο είναι παντελώς παράνομο. Το θέμα μου για την Ουκρανία είναι το εξής. Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας παρακολουθεί κατά κάποιον τρόπο την τελευταία συμφωνία που ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων σχετικά με την παροχή αερίου στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν θέλω που δεν είναι να σκεφτώ ότι αυτή είναι μια εμπορικίστικη προσέγγιση, ότι δεν υπάρχει πίσω από αυτή τη συμφωνία ένα πολιτικό πλαίσιο ένα πλαίσιο που να έχει λάβει υπόψη του και όλες τις προεκτάσεις ε, σε σχέση με την αυτάρκεια ή την διαφοροποίηση σε θέματα ενέργειας τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την Ουκρανία. Ρωτώ λοιπόν, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας πώς παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν θέλουμε η Ουκρανία να εξελιχθεί δημοκρατικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της ε, δημοκρατικής διακυβέρνησης να επικρατήσει αυτή η διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει για την Ουκρανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους ε, αλλοδαπούς μαχητές. Αναφερθήκατε και είπατε ότι είναι ένα είδος ε, τιμωρίας για αυτούς που αποφασίζουν να μεταβούν επί τόπου. Εγώ όμως θα έλεγα ότι είναι ένα λογικό μέτρο με την έννοια της πρόληψης. Όμως και πάλι η προσέγγιση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας ε, πώς ακριβώς αντιμετωπίζει αυτές τις ε, περιπτώσεις των κρατών που τους αφαιρούν την ηθαγένεια στους μαχητές. Αυτό είναι όχι μόνο παράνομο αλλά και αντιπαραγωγικό. Μετατοπίζει την όλη κατάσταση στην περιοχή κατόπιν. Όσον αφορά τις αντιφάσεις ε, της εταιρικής σχέσης με χώρες σημαντικές όπως είναι η Τουρκία, η Σαντική Αραβία ή το Κατάρ υπάρχουν και χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται πάρα πολύ ε, και στηρίζουν το κίνημα ISIS. Εχθές ε, ακούσαμε τον κύριο Μπαρζάνη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος μίλησε για τον έλεγχο ενός δικτύου όπως είναι αυτό του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε συνεργασία με τους Αμερικανούς. Ε, το κάνουμε και τι κάνει η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας τη στιγμή μάλιστα ε, που τα κράτη-μέλη και πολλά άλλα κράτη έχουν ε, συστήματα θεωρήσεων που ξέρετε τελικά αυτά είναι απλά ξέπλυμα χρήματος ε, και εδώ εμπλέκεται και η τρομοκρατία. Και τέλος, ποια είναι η άποψη της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας για το ρόλο του Ιράν στην περιοχή. Διότι το Ιράν είναι, αν θέλετε, η ο βραχίωνας της Σοβιετικής Ένωσης, η ήπια δύναμη που στηρίζει τον Ασάντ. Πήγα στο Ιράν και μίλησα με κάποιους ανθρώπους και μου είπαν ότι δεν θέλουν να σώσουν τον Ασάντ, αλλά δεν επιθυμούν να ενδώσουν σε, στον ακραίο αυτό βραχίωνα το σουνητικό του Ισλάμ που είναι το κίνημα ISIS. Το Ιράν λοιπόν θα μπορούσε να βοηθήσει σε θέματα ασφάλειας και πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για άτυπη συνεργασία με το Ιράν. Όμως και πάλι η πολιτική, Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας πώς ακριβώς διαμορφώνει αυτή τη συνεργασία γιατί ξέρουμε ότι ε, τρέχουν πολύ σημαντικά ε, πράγματα ε, όπως τα θέματα των πυρηνικών. Ο κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπατε χθες, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας έχει συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε λιγάκι για το τι προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, ε, παραδίδονται περισσότερα όπλα από τη Ρωσία, περνάνε από τα σύνορα, παραδίδονται στους αντιστασιακούς, στους τρομοκράτες, πέστε τους όπως θέλετε. Και μπορείτε να μας πείτε μήπως υπάρχει πιο έντονη ε, στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή της Μαριόπολης και μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε περαιτέρω προώθηση των ε, στρατευμάτων της ε, Ρωσίας στη νότια περιοχή. Επανέρχομαι στον μηχανισμό Αθηνά, γιατί είπατε, υπονοήσατε ότι τα κράτη και οι πολίτες θα μπορούσαν να πληρώσουν δύο φορές. Νομίζω ότι αν ε, μεταρρυθμιστεί σωστά ο μηχανισμός Αθηνά, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει αυτό να πληρώνουν δυο φορές τα κράτη-μέλη. Εγώ προσπάθησα να πείσω τις γερμανικές αρχές να δεχθούν αυτή την αρχή της διεύρυνσης και τους είπα ότι τελικά πρώτον θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση, να υπάρξει αποστολή, δηλαδή ομοφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη ότι θέλουν να υπάρξει αποστολή. Και τελικά, αν συμβεί αυτό, τότε γιατί δεν μπορούμε να επιμερίσουμε το κόστος που θα προκύψει. Και θέλω να πω και να πείσω τους Γερμανούς ότι το 22% που είναι το μερίδιό τους, αυτό θα βοηθούσε έτσι ώστε να εμπλακούν και άλλα κράτη-μέλη ανέφερε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Το θέμα της ε, στρατηγικής θαλάσσιας ασφάλειας. Από εκεί προέκυψε συγκεκριμένη αποστολή στον κόλπο της ε, Γουινέας. Οι άνθρωποι... Η Πορτογαλία είχε την υποδομή. Το θέμα είναι όμως ότι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί επαναλαμβάνουν αυτή την αποστολή γιατί κανείς δεν εκλήθη να την καλύψει κατά 100%. Άρα δηλαδή το δικό μου το επιχείρημα είναι να διεξαχθούν συγκεκριμένες συζητήσεις με μεγάλα και μικρά κρατημέλη έτσι ώστε τελικά να υπάρχει μια σωστή αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων και έχοντας κατά νου ότι βεβαίω και πρέπει να εμπλέκονται οι μεγάλοι λόγω της μορφής που έχει λάβει αυτός ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Ο κύριος Κέλλα, μετά υποφαινόμενοι, δεν ξέρω, κάποιος άλλος, αν όχι κλείνει ο κατάλογος των μιλητών. Ο κύριος Κέλλα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε αυτά που είναι μια θετική εξέλιξη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στάθηκε ενωμένη απέναντι στην κρίση της Ουκρανίας. Και πρέπει επίσης ε, να δεχτούμε ότι ο κύριος Πούτινγκ είναι εκείνος που δίνει τον τόνο. Εκείνος ε, δρά και εμείς αντιδρούμε. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Κατά την άποψή σας μέχρι τώρα η αντίδρασή μας ήταν ικανοποιητική κατά τους τελευταίους μήνες γιατί αν ο στρατός της Ουκρανίας ε, θα μπορούσε να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε τον Αύγουστο, τότε νομίζω δεν θα λάμβαν χώρα αυτές οι δίθεν εκλογές. Η Ρωσία είναι εκείνη ε, που χρησιμοποίησε το βαρύ της ε, πυροβολικό, τα βαριά όπλα και αυτά άλλαξαν την κατάσταση και προέκυψε κατάσταση που προέκυψε. Εσείς συμφωνείτε ότι η δική μας αντίδραση ήταν ικανοποιητική το δέχεστε αυτό. Κυρίως ε, στο να ε, εφοδιάσουμε την ε, νόμιμη Ουκρανική κυβέρνηση με όπλα για να αντισταθεί σε αυτή την εισβολή. Και ποιες είναι οι αντίδρασή σας για τα σκάφη Μιστράλ. Αυτό θα παρέκαμπτε την έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αν τελικά δεν χορηγήσουμε όπλα στην νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας και παράλληλα όμως τα κράτη-μέλη να προετοιμάζονται να πουλήσουν πολεμικό σκάφος στον εχθρό. Υπάρχει αυτό το δόγμα της ε, υπεράσπιση συμπατριωτών στο εξωτερικό, δηλαδή χρήση εξωτερικής ε, βίας στο εξωτερικό. Και ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχουν ε, συμπατριώτες ε, για να τους υπερασπιστεί η Ρωσία, η Ρωσία μπορεί να τους δημιουργήσει τεχνητά για να τους υπερασπίσει μετά. Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι χάσαμε την ευκαιρία μήπως να ε, μετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το δόγμα, να το καταργήσουμε, γιατί ξέρετε αυτό αποτελεί τη βάση της συμπεριφοράς της ε, Ρωσίας. Κύριε Πέσβη, θα ήθελα να αναλύσω περαιτέρω το τελευταίο σημείο που έθεσα, να το αλλάξω κάπως, την... να το αντιστρέψω. Εστιάζομαι επί της πολιτικής προσεγγίσεως για την Ουκρανική κρίση και περαιτέρω δράσεις ενδεχομένως και σε άλλες παγωμένες ε, σειράξεις ε, που υπάρχουν στα ανατολικά και ποια είναι η επαρκής δράσης παρατηρώντας ακόμα και τις συζητήσεις μας σε διάφορα βήματα συζητήσεων βλέπουμε ότι ε, εστιαζόμεθα περισσότερο σε τομείς συμφέροντος στον Νότο και την Αφρική εδώ στο Κοινοβούλιο και στη Μέση Ανατολή και ένα μέρος του Κοινοβουλίου εστιάζεται περισσότερο σε απειλές ε, ανατολικά, στην ανατολική γειτονία. Αυτό είναι προφανές. Έχουμε, μάλλον πρέπει, να καταλήξουμε σε σχετικά συμπεράσματα. Λοιπόν, κάθε φορά εγώ θέτω το εξής. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοιου είδους σοβαρές απειλές παντού. Ο κύριος Γκάλερ είχε δίκιο. Έχουμε το δαχτυλίδι της φωτιάς που φλέγεται αντί να έχουμε ασφαλή γειτονιά που θέλαμε να δούμε να υφίσταται όταν θεσπίσαμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας. Θα πρέπει να τονίσουμε εξίσου όλες τις απειλές και να χρησιμοποιήσουμε και τα ίδια πρότυπα όταν υιοθετούμε μέτρα. Θα πρέπει βέβαια να είμαστε και ευέλικτοι. Όμως η ερώτησή μου περιοριζόταν αποκλειστικά στη στατιωτική πτυχή της συνεργασίας με τη Ρωσία ή ενδεχόμενη στατιωτική πτυχή που υφίσταται. Θέλουμε από τη μια σε πολλούς τομείς στην έρευνα σε διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με το διάστημα και σε άλλα προγράμματα θέλουμε πράγματι να δούμε και ποιες είναι οι αμυντικές συνιστώσεις, οι συνιστώσεις ασφαλείας. Και παρόλα αυτά έχουμε συνεργασία με τη Ρωσία που είναι εκείνος που επιτίθεται. Και η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, αυτή τη διαφορά, αυτό το κενό που υπάρχει στην προσέγγιση που ακολουθούμε. Απάντηση, ναι πράγματι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας με τη Ρωσία και στη στατιωτική συνεργασία μας. Είναι, ένα, είναι συνεργασία στις κυρώσεις τρίτου επίπεδου. Έχουμε ακυρώσει κάποιες συνεργασίες στον τομέα υψηλής τεχνολογίας. Και το στρατιωτικό σκάφος, το γαλλικό σκάφος, το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο. Και η Γαλλία βρίσκεται σε δύσκολη θέση ανέβαλαν, νομίζω ανέστειλαν αυτή την απόφαση τους, όμως μπορεί να θέσει ερωτήματα κανείς. Κατά πόσο θα ήταν καλό να γίνει αυτό που πάει να γίνει. Υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις από τις οποίες πρέπει να ξεφύγει η Γαλλία, δεν τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει και το οικονομικό στοιχείο. Όμως έχει τεθεί το ζήτημα. Και η Γαλλία το παλεύει. Για τη στρατιωτική συνεργασία της άλλης πτυχές εντάσσεται στην πολιτική κυρώσεων. Για την ώρα τα κράτη-μέλη πάνω σε αυτά έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν. Και πρέπει να δούμε και τι αποφασίσει το κάθε κράτος ξεχωριστά για τη συνεργασία με τη Ρωσία. Θα μπορούσαμε να θέσουμε εν γέννη ερωτήσεις. Δηλαδή, πώς πρέπει να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια. Και την Παρασκευή ε, ε έγινε όλος προβληματισμός για το θέμα στο πιεσί. E. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ρωσία. Έκανε αυτό που έκανε. Κακή συμπεριφορά. Απ' την άλλη είναι μεγάλος και σημαντικός γείτονας. Δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι δεν υπάρχει. Εκεί είναι. Ήταν αρκετή η αντίδρασή μας επαρκής. Δεν ξέρω. Είχαμε κάποια αντίδραση. Είπα στην αρχή ότι δεν νομίζω ότι υπήρχε δυνατότητα χρήσης στρατιωτική βία. Κάναμε αυτό που ήταν δυνατόν. Υπήρχε δυνατότητα, αλλά όχι πολιτική βούληση από την πλευρά μα, ούτε από πλευρά ΝΑΤΟ. Το θέμα ήταν κυρώσει. Επιβάλαμε αρκετέ κυρώσει. Και πηγαίνουν αρκετά μακριά αυτέ οι κυρώσει αρκούν. Ξέρω ότι κάποιες κυρώσεις πραγματικά πονάνε και έχουν αποτέλεσμα. Αρκεί το αποτέλεσμα. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Συνεχώς παρακολουθούμε την κατάσταση. Προσπαθούμε να αντιδράσουμε. Με διτή προσέγγιση, όπως πάντα. Προσπαθούμε από τη μια να ασκήσουμε πιέσεις και από την άλλη να κρατήσουμε ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας. Αλλά εξελίσσεται η κατάσταση. Η κατάσταση με τις υποτιθέμενες εκλογές στην Ανατολή και εδώ απαντώ στον κύριο Σαφάουζεν, αυτός σου είχε θέσει το ερώτημα. Ναι, κύριο Χάουζερ, χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Όταν έχουμε τη συμφωνία, το πρωτόκολλο του Μίνσκ και τη συμφωνία και η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν κάποια πράγματα. Υπεγράφει. Υπάρχει υπογραφή στο κάτω μέρος της σελίδα. και οι δύο υποσχέθηκαν κάποια πράγματα. Ε, η Ουκρανία έδωσε μεγαλύτερη αυτονομία σε αυτές τις περιοχές. αλλά ξαφνικά όταν επεκράτησε η κατάπαυση του πυρός είδαμε πολλή δραστηριότητα για να κερδίσουν έδαφος οι άλλοι. Παρόλο που δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή μας, μιλούσαμε με κάποιους στατιωτικούς εμπειρογνώμονες που διερευνούν το θέμα αλλά υπήρξε αρκετή δραστηριότητα από την άλλη πλευρά των συνόρων. Τα, τα, τα σύνορα έχουν γίνει πιο διαπερατά. Μπορεί να περνάει κανείς εύκολα τα σύνορα. Ε, στην, στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ έγινε μεγάλη μάχη για τον έλεγχο του αεροδρομίου. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να συνομιλήσει μαζί τους. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε με τα όπλα συνέχεια από ό,τι βλέπω οι άλλοι. Αυτό βλέπουμε οι εκλογές, τι να πω, ήταν σαφές ότι έγιναν εκλογές στην Ουκρανία. Αν θέλει κανείς να εκφράσει τη διαφωνία του, πάντα υπάρχει δημοκρατικός τρόπος να εκφραστεί, καταψηφίζοντας το κόμμα που δεν το αρέσει, αλλά όχι με το να πάρει κανείς τα όπλα του. Τα, τους τελευταίους μήνες που γίνονται οι μάχες είναι σαφές ότι υπήρξαν θέματα και πολλά θύματα και αυτό είναι ατυχές, ατυχέστατο και από τις δύο πλευρές προσπαθούμε και προσπαθούσαμε να σταματήσουμε τις μάχες και είχαμε την κατάπαυση του πυρός. Το πρωτόκολλο του Μίνσκ αποτελούσε τη βάση πρόοδου και βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι το θέμα των συνόρων. Δεν υπάρχει κάποια μετακίνηση, διότι ένα από τα δύο μέρη δεν θέλει να μετακινηθεί. Χρησιμοποιούν την ευκαιρία για να κερδίσουν έδαφος από τον Ουρκανικό στρατό. Στη Μαριούπολη ο βομβαρδισμός υπήρξε, ναι, από ό,τι ξέρουμε. Συνεχίζονται οι μάχες και στον Ντονέτσκ. Υπάρχει ροή όπλων, δεν ξέρω, δεν έχω συγκεκριμένε πληροφορίες, αλλά σίγουρα υπάρχει δραστηριότητα. Και φαίνεται να υπάρχουν και αρκετά προχωρημένα όπλα που προωθούνται στην περιοχή που οι ντόπιοι, ούτε αποκαλούμενοι ντόπιοι, φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά. Μη λησμονούμε αυτό την πτήση MH17 που κατερρίφθη το αεροπλάνο. Δεν το πυροβόλησε μια απλή καραμπίνα, ένα απλό όπλο κάποιου αθώου πολίτη που κυνηγούσε. Πύραυλος το έπληξε, αρκετά περίπλοκο και προθυμένο σύστημα και είναι σαφές ποιος το έκανε αυτό, ποιος κατέρριψε το αεροπλάνο. Υπάρχει τεράστια, τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα σχολεία, για το νερό, δεν μπορεί να κινηθεί κανείς σε ένα πεδίο, σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση και που γίνονται μάχες. Είμαστε έτοιμοι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε. Ήμουν στην Ουκρανία και συναντήθηκα με τον πολιτικό διευθυντή στην Ουκρανία. Ή ε, θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο σε αυτέ τι περιοχέ, να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, να βοηθήσουμε τα σχολεία με δρόμου, ό,τι θέλετε. Έχουμε χρήματα. Αλλά αν δεν έχετε πρόσβαση, τι, τι μπορείτε να κάνετε. Αρχίζουν και πυροβολούν. Πυροβολούν και την αποστολή του ΑΣΕ που συμφωνήθηκε αυτή η αποστολή από όλα τα μέρη. Ε, θα ήταν ανεξάρτητος φορέας. Εκτόξευσαν ε, το τηλεκατευθυνόμενο, όχι, ε, μη επανδρομένο όχημα από την Αυστρία για να παρακολουθήσουμε στα σύνορα, στη συνοριακή περιοχή, μεθοριακή περιοχή. Και το πυροβόλησαν το μη επανδρομένο αυτό αεροπλανάκι, χρησιμοποίησαν τεχνικές ε, για να εκτοχέσουν κάποια τρένα. Αυτή είναι η κατάσταση. Το πρωτόκολλο του Μίνσκ τώρα, τι να πω, οργανώθηκαν αυτές οι εκλογές. Αυτό αντέβαινε τις αρχές του πρωτοκόλλου του Μίνσκ. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε, να δεχτούμε τις εκλογές. Είναι απλούστατο. Αποκαλούνται πρόεδροι βάσει των εκλογών. Κανείς δεν αναγνωρίζει τις εκλογές. Όμως. Ξέρω ότι στηρίζουμε την Ουκρανία ε, ποικιλοτρόπος. Οικονομικά δώσαμε πολλούς πόρους, δίνουμε πόρους. Υπάρχει και επιμερισμός προσπαθειών. Εμείς εξετάζουμε τον τομέα, τον πολιτικό, τον ΝΑΤΟ, εξετάζει τη στρατιωτικό τομέα και βέβαια υπάρχει και στα προγράμματα, υπάρχουν προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας με χώρες του ΝΑΤΟ, όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή, διότι δεν έχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε εκτοξευτές πυράβλων που να στείλουμε στην Ουκρανία. Ξέρω ότι εφαρμόζουν κάποια προγράμματα κράτη-μέλη και ίσως και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει γενική υποστήριξη που παρέχουμε προς την Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια ευρώ διαθέτουμε. Και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορεί να λειτουργεί η Ουκρανία. Είναι μια χώρα που ξεκινά να ανθεί. Και εμεί λησμονούμε όταν βλέπουμε τα επίπεδα ανάπτυξης Πολωνίας και συγκρίνουμε την Πολωνία με την Ουκρανία πριν, πριν από 20 χρόνια κάνουμε τη σύγκριση και να δούμε ποια είναι τα επίπεδα του σήμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια πρόοδος. Ας ελπίσουμε ότι και η Ουκρανία θα μπορέσει να εφαρμόσει μεταρρυθμιστικά προγράμματα, εκδεληφθεί και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη στήριξη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει παράδειγμα η Ουκρανία και να είναι και ελκυστική ε, χώρα για τους πολίτες. Για το μηχανισμό Αθήνα συμφωνώ κύριε Γκάλερ με την ανάλυση σας το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι κάποιες χώρες, να μην κατονομάσω συγκεκριμένες, κάποια χώρα λέει ναι είμαι μεγάλη χώρα όμως, είμαι πιθανότατα μία από τις χώρες, λίγες χώρες που μπορεί να διαθέσει επαρκές στατιωτικό υλικό και εξοπλισμό αν, θέλει, αν πρέπει να συμβάλλω και στο κοινό κόστος παραπάνω οικονομικά σημαίνει ότι πληρώνω διπλά. Αυτή τη λογική ακολουθούν. Είναι κάπως παράλογο, αυτή τη λογική ακολουθούν όμως. Και ίσως είναι εύκολο να βρει κανείς αντεπιχειρήματα αλλά είναι ίσως πιο είναι θεωρητικά, θεολογικά θα έλεγα επιχειρήματα. Θεωρούν ότι δεν είναι καλό να αναπτυχθεί πολύ κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Ό,τι πάει προς, προς αύξηση της ευρωπαϊκής κοινο... ε, ε, πολιτικής τους βρίσκει αντιθέτους. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουμε και χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ο ρόλος του Ιράν, σημαντικότατο θέμα αλλάζει η εικόνα. Διότι το Ιράν Βεβαίω, και παίζει κάποιο ρόλο στη Συρία, στη σχέση του με τη Χεσμπολά. Από την άλλη όμως πλευρά βλέπουμε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Έχουμε ε, την εξέγερση των Σούνι και οι Σούνι και οι Σουνίτες, με συγχωρείτε, οι Σουνίτες και οι Σίτες, ε, γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματά μας. Επίσης ε, μιλάμε με το Ιράν γιατί το Ιράν είναι μια σημαντική χώρα στην περιοχή και τώρα αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν είναι εύκολο βέβαια και όλα αυτά έχουν σχέση και με τις ε, συζητήσεις ε, για τα πυρηνικά όπλα. Ε, προσπαθούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά, αλλά είναι πολιτικά συνδεμένα μεταξύ τους. Πάντως, 24 Νοεμβρίου θα υπάρξει μια συμφωνία Μπορείτε να φανταστείτε τις ε, συνέπειες αυτής της συμφωνίας και στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά πετρελαίου θα είναι τελείως διαφορετική γιατί οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να πέσουν ε, και τότε η Ρωσία θα αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τις ε, στρατηγικές αλλαγές στις οποίες έχουμε μπλακεί. Ναι, πρέπει να μιλάμε με το Ιράν και με το Κατάρ με τη Σαουδική Αραβία παρά το ρόλο που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν. Και ξέρετε κάποια στιγμή όταν ε, ένα μεγάλο κράτος λέει ότι ε, θα ε, κατευθύνει, θα χειρίσει την κατάσταση από το παρασκήνιο, τότε δημιουργείται ένα μεγάλο κενό και το κενό δεν παραμένει για πολύ καιρό, αυτό πληρούται. Αυτό συνέβη. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το ότι το Κατάρ, τα Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία όλοι ε, εντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια κατά του ISIS. Όσον αφορά το θέμα των αλλοδαπών μαχητών ε, και την, εθνική, την ε, ηθαγένεια. Ε, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα των Υπουργών ε, Εξωτερικών. Αλλά έχουμε μια κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών και εκεί θα εξετάσουμε την στρατηγική ε, από το πρίσμα της εξωτερικής ασφάλειας. Τι μπορούμε να κάνουμε με τους εταίρους, με την Τουρκία και με άλλους και επίσης με τους συναντέλφους μας από το εσωτερικό μέτω. Και εκεί ε, βλέπουμε ότι έχουν αφαιρεθεί διαβατήρια για να μην ε, φύγουν οι άνθρωποι, αλλά βλέπουμε ποιες είναι οι συνέπειες. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία για το αέριο, δεν είναι στη δική μας την ε, ημερήσια διάταξη, αλλά και αυτό εντάσσεται στα ευρύτερα θέματα. Υπάρχει ένα είδο αναγκαιότητα, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συμφωνία γιατί έρχεται ο χειμώνα. Όμω αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική ατζέντα ε, περί Ουκρανίας. Εμείς στηρίζουμε την Ουκρανία αλλά πρέπει ε, να τους στηρίξουμε και να αποκτήσουν το απαραίτητο αέριο για να περάσουν το χειμώνο. Αυτά ε, μέσα στο πολιτικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικά και νομίζω όλοι τα χαιρέτησαν στο πλαίσιο της ε, Επιτροπής Πολιτικής Ασφαλείας αλλά και στο πλαίσιο της Κορεπέρ. Νομίζω ότι μίλησα, μάλλον απάντησα για το θέμα του στρατιωτικού εξοπλισμού και νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρέσβη, θα συνεχίσουμε αυτή τη βιτή προσέγγιση αφενός λαμβάνουμε υπόψη μας τις εξελίξεις ε, της ε, ΚΠΑ και από την άλλη θα αξιολογήσουμε τις ε, προκλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και θα αναζητήσουμε ικανοποιητικές ε, απαντήσεις σε επίπεδο οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη που ήρθατε. Ένα λεπτό διάλειμμα για να ε, αναδιαταχθούμε και θα ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα. Ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε παρακαλώ. We go to the next point of... Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι το θέμα της ασφάλειας και των πτυχών άμυνας σε, δύο, σε σχέση με δύο προγράμματα, το Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο. Γαλιλαίο και Κοπέρνικους. Με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να, να παρουσιάσω τους τρεις συμμετέχοντες, επαΐοντες, πραγματογνώμονες. Πρώτα τον κύριο Φρανκ Ασμπεκ, που είναι ο κύριος σύμβουλος αρμόδιος για θέματα πολιτικής, διαστήματος και ασφάλειας μέσα στο πλαίσιο της ΕΕΔ, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και υπό αυτή την ιδιότητα του ξεχωριστά που θα σας αναφέρει τα σχετικά και δεύτερον έχουμε δύο κυρίους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόντες, τον κύριο Πολ Φλαμόν και τον κύριο Μάουρο Φακίνη, που είναι και οι δύο εμπλέκονται σε θέματα που αφορούν και το Γαλιλαίο και, τον, και το Κοπέρνικους. Πρώτα έχετε εσείς τον λόγο κύριε Άσπεκ, παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το ότι με προσκαλέσατε σήμερα εδώ ενώπιον σας για να ομιλήσω για ένα θέμα που έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία και σπουδαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πτυχές ασφάλειας όσον αφορά τη διαστημική πολιτική. Και η διαστημική πολιτική ραγδαία αναπτύσσεται με δραματικό τρόπο ως θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι εμπλέκονται και θέματα άμυνας και ασφάλειας φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πτυχές ασφάλειας πάντα ήταν αδιάρρηκτες όσον αφορά το διάστημα και τη διαστημική. Σε μεγάλο βαθμό φυσικά <clears throat> στο διάστημα και τη διαστημική και την ειρήνη και την ισορροπία και ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και όλο και περισσότερο η διαστημική τεχνολογία στις περισσότερες φορές, περισσότερες φορές είναι διτής, διπλής χρήσης και οι διαστημικές εφαρμογές ε, είναι διπλής χρήσης και εφαρμογής ε, εφαρμογές. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει πάντα να θυμόμαστε όταν κάνουμε λόγο για θέματα διαστήματος και διαστημική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το, τη διαστημική και το διάστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αργά ε, κατέληξε σε αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μια κίνηση κατά, την, ε, κατά το τέλος του ψυχρού πολέμου ατομικά επιμέρους για τα κράτη-μέλη και συλλογικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν κατά τη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας 90 ξεκίνησε μέσα στο πλαίσιο της ε, Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Ευρώπη να αναπτύσσει αυτές τις ε, δράσεις, δημιούργησε το ε, δορυφορικό κέντρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992. Στόχος ήταν να υποστηρίζονται οι αποφάσεις ε, που λαμβανόντουσαν και θα λαμβανόντουσαν όσον αφορά την ασφάλεια και θέματα ασφάλειας και άμυνας στο διάστημα. Και μέσα στο πλαίσιο των ε, στόχων και καθηκόντων Πέτερσμποργκ 1992 ανθρωπιστική βοήθεια, διασφάλιση Ειρηνη και συντονισμό ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά ειρηνευτικέ πρωτοβουλίε και δράσει. Αν θέλουμε πολιτικές αποφάσεις να εφαρμόζονται και να λαμβάνονται υπόψη στα θέματα ασφάλειας, πρέπει έγκαιρα να έχουμε πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα. Καλές πληροφορίες δεν διασφαλίζουν τις καλές αποφάσεις. Όμως κακές πληροφορίες διασφαλίζουν κακές αποφάσεις. Και γι' αυτό ήταν ένα αυτό για τα κράτη της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνώρισαν ότι η δορυφορική ανείχνευση και αναγνώριση ήταν θεμελιώδες στοιχείο για μια ορθή πολιτική ασφάλεια ασφάλειας Όλα τα κράτη θα έπρεπε σε, σε μια κοινή βάση ως πλατφόρμα να λαμβάνουν στοιχεία για τις αποφάσεις τους και έτσι με βάση το δυναμικό των κρατών μελών να μπορούν να δράσουν λαμβάνοντας και μια κοινή απόφαση για κοινή δράση εν καιρό. Αυτό το θέμα δεν έχει αλλάξει, αυτό το πλαίσιο δεν άλλαξε όταν εντάχθηκε το δορυφορικό κέντρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέος οργανισμός το 2002 για πολιτικούς οργανισμούς όπως η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση το δορυφορικό κέντρο προσφέρει σαφώς προτερήματα όσον αφορά πληροφορίες για περιοχές κρίσης ή σειράξεων όταν χρειαζόμαστε τέτοιες πληροφορίες από εκεί παγκόσμια οικουμενική προσπέλαση και πρόσβαση που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να αποκτηθούν λόγω του απόμακρου χαρακτήρα τους, λόγω των υποδομών κτλ. Δορυφορική παρατήρηση δίνει άμεση πρόσβαση. Μέσα σε λίγες μέρες, πολλές φορές μέσα σε λίγες ώρες. Πρώτες πληροφορίες μπορούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να διατίθενται ασφαλώς ασφαλή πρόσβαση για παράδειγμα. Για παράδειγμα, αν η προσπελασιμότητα δεν είναι δυνατόν να διασφαλίζεται από τους συμμετέχοντες σε μια σύραξη, σε μια περιοχή, σημαντικό είναι το δορυφορική, η δορυφορική ανείχνευση με πλήρη σεβασμό των διατάξεων του διεθνούς δικαίου να μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να δράσουμε, χωρίς να χρειάζεται να διαβουλευτούμε με κανέναν ή να προηγηθεί κάτι άλλο. Για παράδειγμα, παρουσία παρατηρητών ε, για ανθρωπιστικές δράσεις πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί επιτόπου. Οι δορυφορικές ε, απεικονίσεις και εικόνες και πληροφορίες μας δίνουν αυτά τα στοιχεία κατά πόσον δηλαδή κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό ή όχι. Αυτές οι πληροφορίες εύκολα μπορούν να διαχυθούν και να αποτελούν αντικείμενο κοινού προβληματισμού για τα κράτη-μέλη. Το δορυφορικό κέντρο διαδραμάτισε αυτό το ρόλο του τα τελευταία 20 χρόνια και είναι ένα ανεκτήμητο στοιχείο για την ε, λήψη αποφάσεων και προετοιμασία αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ας περάσω στον Κοπέρνικο τώρα και τη σπουδαιότητά του για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Το Κοπέρνικος φυσικά έχει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στο να επιτύχει αυτόνομες ε, δράσεις όσον αφορά την παρατήρηση της, ε, των, ε, όσων τεκταίνονται επιγείως. Ένας από τους στόχους είναι να αντιδράσουμε στην άμεση ανάγκη των αρμόδιων για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής με βάση τις εικόνες από δορυφόρους και τα στοιχεία μεσοδορυφόρων. Όταν ως GMES ε, συνελήφθη η προσέγγιση αυτή η ιδέα του Κοπέρνικους ήταν ένα ε, κέντρο οικουμενικό για θέματα ασφάλειας. Άλλαξε αμέσως αυτό σε πολύ μικρό διάστημα για τις παρατηρήσεις περιβάλλοντος και ασφάλειας. Αυτό δείχνει ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος, θεμάτων περιβάλλοντος, έχει επιπτώσει στα θέματα ασφάλειας. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κάνουν λόγο για το GNSS, δηλαδή για το σύστημα δορυφορικών παρατηρήσεων και δορυφορικού εντοπισμού στην εισαγωγή μου ε, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, υπάρχουν έξι κέντρα για ε, το περιβάλλον, τις ατμοσφαιρικές αλλαγές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις υπηρεσίες που έχουν σημασία για τις συζητήσεις μας σήμερα για την ε, κατεπίγουσα διαχείριση περιπτώσεων και για την διαχείριση περιπτώσεων ασφάλειας. Η υπηρεσία ασφάλειας έχει τρία στοιχεία. υποστήριξη της εξωτερικής δράσης το ένα το άλλο είναι η εποπτεία συνόρων. Το άλλο είναι η ναυτιλιακή, η ναυτική εποπτεία. Έχουμε ήδη στην έκθεση που υπευλήθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά το Δεκέμβριο 2013 τα συναφή και δηλώσαμε ότι, δηλώθηκε ότι η εξωτερική υπηρεσία εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιεί το Κοπέρνικο στις εξωτερικές δράσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα εργασίας του Κοπέρνικους προβλέπει ότι το δορυφορικό κέντρο θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και στις μελλοντικές υπηρεσίες και δράσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δορυφορικό κέντρο έχει μακρά πείρα και εμπειρία στην αντιμετώπιση απορρίτων και διαβαθμισμένων στοιχείων για να υποστηρίζεται η διαδικασία λήψης απόφασης στην κοινή εξωτερική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είναι σημαντική η δράση του για να διασφαλίσετε μια συντονισμένη δράση και προσέγγιση όσον αφορά καθήκοντα που αφορούν το Κοπέρνικους αφενός μέσα στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής και την χρήση του δορυφορικού κέντρου αφετέρου που πρέπει να διασφαλίζεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια οπωσδήποτε. Και για αυτούς τους λόγους το δορυφορικό αυτό κέντρο ήδη λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προλειτουργικές υπηρεσίες που διασφαλίστηκαν μέχρι σήμερα προετοιμάζοντας, προλιένοντας την λειτουργική τους φάση. Το χαρτοφυλάκιο της υπηρεσίας αυτής καθορίστηκε όσον αφορά το φάσμα, το εύρος του και είναι ευρύτατο το φάσμα αυτό από την διασφάλιση βασικών χαρτών μέχρι την εποπτεία και παρακολούθηση προσφυγικών ε, καταβλισμών την εξόριξη ορυκτών και μεταλλευμάτων, την αξιολόγηση των καταστάσεων οδικών δικτύων και δρόμων και των υποδομών, το κέντρο ε, αποτίμησης ε, σειράξεων και συγκρούσεων, η παρακολούθηση παράνομων καλλιεργειών σε τομείς όπου καλλιεργούνται τέτοιες παράνομες καλλιέργειες, για παράδειγμα για την παραγωγή ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Είναι όριμη λειτουργικά αυτή η υπηρεσία. Ωστόσο πρέπει να διασφαλιστεί σωστή διαχείριση και διακυβέρνηση. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το νομικό πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας Λαμβάνοντα υπόψη ότι το δορυφορικό κέντρο είναι μια υπηρεσία τη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, με παρουσία τη ΥΠΑ της εκπροσώπου και τη υπηρεσία εξωτερική δράση για τι λειτουργικέ δράσει, καθώ επίση και την πολιτική επιτροπή και πολιτική ασφάλεια που έχει τη συνολική εποπτεία. Θα συνεισφέρει το δορυφορικό κέντρο σε άλλε δράσει των, από πλευρά Κοπέρνικου, ιδιαίτερα για την εποπτεία συνόρων, παρακολούθηση συνόρων. Από τότε που ξεκίνησε αυτό το κοινό και αυτό, το κέντρο εμπλέκεται στον καθορισμό και λειτουργία των ε, μεθοριακών και, ε, και συνοριακών ε, παρακολουθήσεων. Η λειτουργία μεταξύ αυτού του κέντρου και Frontex βρίσκεται υπό προπαρασκευή. Δείχνει ποιες συνέργειες μπορούν να υπάρξουν μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών ασφάλειας που συζητήθηκαν σήμερα το πρωί νωρίτερα εδώ στο, στο δικό σας όργανο καθώς επίσης επιπρόσθετα τέτοια συνεργασία οδηγεί στο να αποφεύγεται επικάλυψη προσπαθειών και δράσεων από πλευράς οργανισμών και υπηρεσιών. Η ίδια συνεργασία αναζητούμε να διασφαλιστεί όσον αφορά την παρακολούθηση ναυτιλιακών θεμάτων, ναυτικών θεμάτων ε, και θεμάτων της θάλασσας ε, και της εποπτείας. Ε. Τη θαλάσσια εποπτεία. Τώρα να μιλήσω για τα θέματα αυτά όσον αφορά το Γαλιλαίο και την ε, συνολική ε, δράση που παρέχεται επικουρικά. Αποστέλλονται μηνύματα στους χρήστε, ε, δίνοντας στίγματα και πληροφορίες συναφή. Η σπουδαιότητα αυτή της τεχνολογία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να υπερεκτιμηθεί οι μεταφορές, ε, οι, ε, τα θέματα ανεφοδιασμού, η αλυσίδα ανεφοδιασμού, η, ε, τα θέματα ενέργειας, γεωργίας και άλλα πολλά εξαρτώνται από την σαφή, τον σαφή προσδιορισμό στιγμάτων έγκαιρα και όσον αφορά και την αυτιλία τα κράτη συνεργάζονται για την διασφάλιση αυτού του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΠΑ, η Κίνα, η Ινδία ε, και η Ιαπωνία συμμετέχουν. Το δορυφορικό σύστημα Γαλιλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίζει την ευρωπαϊκή αυτονομία, ώστε να εγγυόμεθα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, υπηρεσίες υπό ευρωπαϊκό έλεγχο και διαχείριση είναι και υπό πολιτικό έλεγχο και έτσι διασφαλίζεται η αναγκαία υποδομή για τις λειτουργίες από τις οποίες εξαρτώνται οι κοινωνίες μας. Μια και υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών και για τον εντοπισμό στίγματος και για την χρονική αλληλουχία και έγκαιρο διασφαλισμό, αυτό μπορεί να διασφαλίσει ε, πολλά προτερήματα. Έχει λοιπόν μια πολύ σημαντική συνιστόσα όσον αφορά, παράμετρο όσον αφορά την ασφάλεια και για τις PRS, Public Regulated Services, ε, δημόσια διασφαλιζόμενες ε, υπηρεσίες από πλευράς ε, των κυβερνήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο ποιότητας και συνέχεια. Ασφαλή μηνύματα ηλεκτρονικά διασφαλίζονται που μεταφέρονται, διαβιβάζονται. Θα περιορίζεται η διαβίβαση στα κράτη-μέλη και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέλλον όμως και τρίτα κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ε, δημόσια διασφαλιζόμενη υπηρεσία υπό το πλαίσιο συμφωνιών που πρέπει να συναυθούν όμως. Έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία υπό πολιτική και στρατηγική πτυχή. Για θέματα ασφάλειας ε, και άμυνας ε, θα υπάρχει στενότατος έλεγχος από πλευράς μας η προσέγγιση στα ακριβή στίγματα ναυτιλίας έχει τεράστια σημασία για τις ε, ένοπλες δυνάμεις και δυνάμεις ασφάλειας ε, και επιβολής του νόμου όπως αστυνομικές δυνάμεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοια μηνύματα και από τα, ε, τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών αν αποφασίσουν να το πράξουν. Και αυτό φυσικά θα ε, οδηγήσει ε, στο να απεμπλακούν αυτές οι ένοπλες δυνάμεις από την χρήση του αμερικανικού συστήματος ε, δορυφορικής ναυτιλίας και εντοπισμού στίγματος. Και αυτό είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για μας. Η ύπαρξη του συστήματος GNSS μπορεί να οδηγήσει στο να αντιμετωπιστούν πιθανέ απειλέ εν δυνάμει που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να προέρχονται από μια εχθρική δύναμη τέτοιου είδου απειλέ, όπω από μια τρομοκρατική ομάδα ή συμμορία που μπορεί να χρησιμοποιήσει να καταχραστεί τέτοιων μηνυμάτων ώστε να μπορέσουν να καθοδηγήσουν μη επανδρομένα αεροσκάφη, να οδηγήσουν στην έκρηξη εκρηκτικών. Μπορεί εχθρικέ δυνάμει να προσπαθήσουν να αδρανοποιήσουν αυτό το ίδιο δορυφό δορυφορικό σύστημα ώστε να μην το χρησιμοποιούν οι χρήστες. Παράδειγμα, με επιθέσεις επίγειων σταθμών ή υποδομών ή χρησιμοποιώντας επίσης και δορυφορικό δυναμικό κατά του δορυφορικού συστήματος Γαλιλαίου. Τέτοιου είδους απειλές συμπεριλαμβάνουν παρεμβάσεις, παρεμβολές στα συστήματα συχνοτήτων, το spoofing επίσης ή κυβερνοεπιθέσεις και οι συνέπειες αυτών των ε, ε, προβλημάτων ε, για το Γαλιλαίο θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη εμβέλεια, να δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Αν μια τέτοια απειλή αναδύεται, έχει κέρια σημασία οι αναγκαίες αποφάσεις να μπορούν άμεσα να ληφθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγες ώρες όλες όλες ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η απειλή και η απάντηση, η αντίδραση θα μπορούσε να είναι η χρονική ή τοπική τροποποίηση των μηνυμάτων των ε, ε, διαβιβάσεων Γαλιλαίου ώστε να είναι μόνο διαθέσιμα σε εγκεκριμένους χρήστες. Μια τέτοια απόφαση καθώς εμπλέκει την ασφάλεια των κρατών μελών και θέματα κριτικών υποδομών το Συμβούλιο το 2004 υιοθέτησε και τον Ιούλιο και πάλι το 2014 ενέκρινε μια απόφαση που ε, διευθετεί τα θέματα αυτά λήψης απόφασης προς το Συμβούλιο. Σε κατεπίγουσες περιπτώσεις η ύπατη εκπρόσωπος ή ο ύπατος εκπρόσωπος θα πρέπει να λαμβάνει αυτή την ενδιάμεση απόφαση που μπορεί να τροποποιείται μετά στη συνέχεια από το Συμβούλιο. Επιτρέψτε, με, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αναφέροντας δύο λόγια για το περιβάλλον δι, ε, διαστημικής μέσα στο οποίο λειτουργούν όλα αυτά. Σήμερα το διάστημα είναι πραγματικά υποσυμφόρηση υπό, από υπερβολικά πολλούς δορυφόρους ε, μέσω της πολιτικής που ακολουθήθηκε και από τη ΣΥΠΑ. Η κατάσταση επιδεινώνεται και έτσι όλο και περισσότερες απειλές ε, και κίνδυνοι αναδύονται. Λοιπόν, παρέμβαση με τους και φυσική καταστροφή μπορεί με αντιδορυφορικά συστήματα και θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν χώρες που αναπτύσσουν και δοκιμάζουν τέτοιου είδους ε, οπλικά συστήματα. Άλλοι κίνδυνοι όπως ηλιακές επιρροές, ε, μαγνητικές καταιγίδε, ε, διάφορες εκρήξεις του ηλίου, ηλιακές εκρήξεις, ηλιακό κλίμα αποκαλείται αυτό καμιά φορά, διάφορα κομμάτια, ρήματα από το διάστημα, ε, δυσλειτουργίες των δορυφορικών συστημάτων κλπ. Λοιπόν, αυτά τα απορρίμματα του διαστήματος ε, συμβάλλουν κατά πολύ στο, στη συμφόρηση του διαστήματος και αυτό προσέχεται όλος ιδιαίτερος από τη διεθνή κοινότητα σαν φαινόμενο. 15.000 τεμάχια πορυμάτων μεγαλύτερα των 5 εκατοστών είναι σε τροχιά γύρω από τη γη και περίπου 600.000 κομμάτια μεγαλύτερα από το 1 εκατοστό ε, είναι σε τροχιά και έχουν κινητική ενέργεια ένα, γραμμάριο, ένα κομμάτι ενός γραμμαρίου ε, με την ταχύτητα που κινείται έχει μεγάλη κινητική ενέργεια. Αντιστοιχεί στην ενέργεια που ελευθερώνεται από μια έκρηξη χειροβομβίδας για να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Έχουν καταστραφεί σε τροχιά δορυφόροι. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε μόνο τη σύγκρουση του 2009 ανάμεσα στο δορυφόρο Κόσμος 2251 και το, με τον Iridium 33 δημιούργησε περίπου 600 τέτοια κομμάτια θραύσματα. Τον Ιανουάριο του 2007 έγινε μια δοκιμή των Κινέζων συστήματος κατά δορυφόρου και δημιούργησε 2.500 τεμάχια από τέτοια συντρίμια. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις, τη μία την ανέφερα ήδη, όταν αναφέρθηκα στον Γαλιλαίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει επιχειρησιακές διαδικασίες για να αντιδρά αν οι δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόβλημα, κινδυνεύσουν. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει την διαστημική της ευαισθητοποίηση. Όπως θα γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έλαβαν απόφαση να δημιουργήσουν ε, ένα πρόγραμμα για στήριξη και εποπτεία του διαστήματος βάσει ε, μηχανισμών και ε, υποδομών που έχουν τα κράτη-μέλη. Οι προπολογισμοί για το Γαλλιό και τον Κοπέρνικο συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του όλου προγράμματος. Το κέντρο, το δορυφορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξει σημαντικό ρόλο θα μπορεί ε, να είναι ένα ε, σημείο συγκέντρωση στοιχείων που ατεδεθέτει στους χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και ανάλογα με το τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι χρήστες. Μετά χρειάζεται και πολιτική πρωτοβουλία ε, την οποία θα ήθελα να αναφέρω και θα είναι το τρίτο βασικό πρόγραμμα ε, της διαστημικής πολιτικής Ευρώπης. Δηλαδή πρόταση για διεθνή διοντολογικό κώδικα για διαστημικές δραστηριότητε. Αυτός ο κώδικας θα πρέπει να στηρίζει την ασφάλεια και βιωσιμότητα του διαστήματος, ε, δημιουργεί εμπιστοσύνη και διαφάνεια καλύπτει και το θέμα της μειώσεως των, αυτών των, συντριμίων, των αυτών των συντριμιών του διαστήματος. Έχουμε ξεκινήσει διαβουλεύσεις και έχουν συμμετάσχει πάνω από 90 κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Ξεκίνησε τον ΟΗΕ συζήτηση ε, και ελπίζουμε ότι όλη η διαδικασία θα μπορέσει τελικά να καταλήξει κάπου θετικά και στο εγγύς ε, μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άσπεκ. Ο κύριος Πολ Φλαμό έχει το λόγο. Κυρία Προέδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να έρθω και να αναφερθώ στην πρόοδο των προγραμμάτων, των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης Πιστεύω ότι αποδεικνύει πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σα υπενθυμίσω ότι ο επίτροπός μου, ο τότε επίτροπός μου, η κυρία Νέλη Φερόση ήρθε να κάνει μια έκθεση προόδου για τα συστήματα πλοήγησης στην Επιτροπή Ήτρε ε, τον μήνα Σεπτέμβριο. Μίλησα, αναφέρθηκα σε δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, διότι πολύ συχνά τα ε, ταυτοποιούμε αυτά τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης με το Γαλιλαίο και μόνο με το Γαλιλαίο. Ε, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ότι έχουμε ήδη ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργικό, το EGNOS, το οποίο βασίζεται στο GPS αλλά βετιώνει τα χαρακτηριστικά του GPS στην ευρωπαϊκή επικράτεια και αυτό το σύστημα λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και χρησιμοποιείται βασικά στον τομέα της ε, αεροναυτικής, τον αεροναυτικό τομέα και οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι διότι μεγάλος αριθμός διαδικασιών προσγείωσης σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ε, πολλαπλασιάζονται το έγνος ήδη έχει αποδείξει τη δυνατότητα που έχουν οι διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς, η Ευρωπαϊκός Διαστημικός Φορέας ε, και διάφοροι βιομηχανικοί φορείς να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα μεγάλης εμβέλειας στην ε, δορυφορική πλοήγηση. Όπως ε, πριν από δύο λεπτά είπε ο κύριος Ασμπέκ, η δορυφορική πλοήγηση είναι σημαντικότατη. 7% του ΑΕΠ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από την δορυφορική πλοήγηση. Όχι μόνο για θέματα ε, στίγματος, εντοπισμού στίγματος, αλλά και για συγχρονισμό σε πολλούς τομείς, όπως το ενεργειακό τομέα, οικονομικών συναλλαγών ή κινητής ε, τηλεφωνίας. Πού βρισκόμαστε λοιπόν όσον αφορά το Γαλιλαίο και το Έγνος. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε αρχικά ότι χάρη στο νομοθέτη ε, έχουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης και μια σταθερή χρηματοδότηση για το παρόν πλαίσιο το επταετές. Πιστεύω ότι αυτό το εκτιμούμε πολύ, διότι επιτρέπεται έτσι σε όλους τους φορείς δορυφορικής πλοήγης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται σε ένα πλαίσιο σταθερό και έτσι μπορούν να συγκεντρωθούν στο έργο τους για να λειτουργήσουν οι υποδομές τους. Μια υπενθύμηση λεπτομέρειας όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Καταρχάς γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαχειρίζεται το πρόγραμμα και έχει ευθύνη απέναντι σε εσά ε, στο Κοινοβούλιο και έναντι του Συμβουλίου. Να γνωρίζετε επίσης ότι όλες οι υποδομές του Γαλιλαίος και του Έγνος ε, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται σε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε διακυβερνητική υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που είναι το, το τεχνικό μας σκέλος, μας βοηθά να αναπτύσσουμε και να λειτουργούμε αυτά τα συστήματα. Και μετά, όπως γνωρίζετε, εδώ και κάποια χρόνια δημιουργήσαμε έναν οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιφορτίζεται με την εκμετάλλευση του συστήματος, των συστημάτων. Η ΖΕΣΑ είναι ο φορέας αυτός, εδρεύει στην Πράγα, η GSA και εκμεταλλεύεται το έγνος και σε κάποια χρόνια θα εκμεταλλεύεται και το Γαλιλαίος. Το Γαλιλαίος. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήματος. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα τμήματα στο Γαλιλαίος. Μία υποδομή ε, στο έδαφος και μία υποδομή στο διάστημα. Πολύ συχνά οι άνθρωποι δεν βλέπουν παρά μόνο το ορατό κομμάτι του παγωβάνου που, παγωβούνου που είναι ε, οι ανθρωποι δεν βλεπουν παρα μονο το ορατο κομματι του που παγωβουνου που ειναι οι δορυφοροι 90% του συστήματος είναι στις ε, υποδομές της γης. Ε, η υποδομή αυτή είναι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε διεθνή διάσταση σημαντική μάλιστα. Έχουμε σταθμού στο Βόρειο Πόλο, στο Νότιο Πόλο, στα, στην Πολυνησία, πάντα σε επικράτεια που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δύο μεγάλα τμήματα της υποδομής του Γαλιλαίος είναι τα κέντρα ελέγχου και τα κέντρα ασφαλείας. Έχουμε δύο κέντρα ελέγχου και δύο κέντρα ασφαλείας τα οποία τα κέντρα ελέγχου κατευθύνουν τους δορυφόρους και κατασκευάζουν τα μηνύματα πλοήγησης και τα τμήματα ασφαλείας εξασφαλίζουν κάθε πρόβλημα ασφαλείας να παραμένει υπό έλεγχο και ε, ε καλύπτουν και το Γαλιλαίος όπως σας είπα. Αυτά όσον αφορά τις ε, υποδομές στο έδαφος. Για τις υποδομές στο διάστημα ε, θα γνωρίζετε ότι ήδη χάρη στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος εδώ και κάποια χρόνια έχουμε εκτοξεύσει τέσσερις δορυφόρους που μας επέτρεψαν να κάνουν πολλές δοκιμές όσον αφορά το σύστημα και την όλη σύλληψη του συστήματος. Από το 2013 διαπιστώσαμε ότι η σύλληψη του συστήματος είναι έξοχη διότι το 2013 καταφέραμε για πρώτη φορά να υπολογίσουμε τις θέσεις στο έδαφος χάρη αποκλειστικά σε αυτούς τους τέσσερις δορυφόρους. Το σύστημα λειτουργήσε και παραπάνω τις ελπίδες μας, διότι η ακρίβεια της, του εντοπισμού στίγματος ξεπερνούσε ακόμα και αυτό που ήθελαν οι μηχανικοί αρχικά. Χάρη σε ατομικά ρολόγια πάνω στους δορυφόρους, στους δορυφόρους που είναι εξαιρετικά ακριβοί. Ε, εκτοψέξαμε τον Αύγουστο δύο δορυφόρους και θα μίλησε δύο λεπτά για αυτούς. Και μετά επίσης έχουμε δρομολογήσει την παραγωγή 20 δορυφόρων από τη γερμανική εταιρεία OHB. Οι δύο δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν τον Αύγουστο τοποθετήθηκαν σε τροχιά που δεν ήταν η προβλεπόμενη. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος εργάζεται προσπαθώντας να διορθώσει την κατάσταση, να επανατοποθετήσει τους δορυφόρους και σήμερα, ακριβώς σήμερα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ξεκίνησε κάποιες επιχειρήσεις με αυτούς τους δορυφόρους, γιατί αυτοί οι δορυφόροι παρά το γεγονός ότι είναι σε κακή τροχιά ε, είναι υπό πλήρη έλεγχο. Σήμερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ξεκινά τη μετακίνηση των δορυφόρων από αυτή την τροχιά για να τους προσεγγίσει στην τροχιά στην οποία θα έπρεπε να είναι ευθύς εξ αρχής. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να, να πετύχουμε τον αρχικό, την αρχική τροχιά αλλά θα πλησιάσουμε αρκετά και έχουν, θα ξεκινήσουν δοκιμές πάνω στους δύο δορυφόρους το Δεκέμβριο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συναγάγουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και του χρόνου τον Ιανουάριο θα δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα ή όχι να εκμεταλλευτούμε επιχειρησιακά, λειτουργικά αυτούς τους δύο δορυφόρους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας της διάρκειας ζωής που έχουν. Για τους 20 δορυφόρους που παράγονται από τη γερμανική εταιρεία OHB θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα τους εκτοξεύσουμε χάρη σε εκτοξευτές εκτοξευτήρες που που είναι σε σύμβαση με την Ariane Σπάς. Έχουμε τέσσερις σογιούς, ε, εκτοξευτήρες σογιούς. Ο κάθε εκτοξευτήρας σογιούς επιτρέπει την εκτόξευση δύο δορυφόρων κάθε φορά και έχουμε και σύμβαση με την Ariane Εσπάς για τρεις εκτοξευτές Ariane 5. Κάθε πύραυλος Αριάν 5 επιτρέπει την εκτόξευση τεσσάρων δορυφόρων ταυτόχρονα. Ε, υπάρχει και ένα σημαντικότατο τμήμα των εργασιών μας που επικεντρώνεται επί των χρηστών γιατί να δημιουργήσουμε την υποδομή αν δεν βασιζόμαστε στις ανάγκες των ε, χρηστών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε ένα κέντρο υπηρεσίας όπως το αποκαλούμε, εστιακό ε, σημείο για τους χρήστες και αυτά τα κέντρα υπηρεσίας βρίσκονται στη Μαδρίτη και ήδη ε, εν μέρη λειτουργεί το κέντρο αυτό στην Μαδρίτη. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ούτως ώστε να δημιουργήσουμε εφαρμογές που θα γίνουν δυνατές χάρη στο Γαλιλαίος αλλά και χάρη και στο έγνος. Και εν συνεχεία η υπηρεσία μας της Πράγας, η GSA, συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές δεκτών πλοήγησης δορυφορικής στον κόσμο και είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον τους κατασκευαστές δεκτών και έχουμε κάνει και δοκιμές στα εργαστήρια που λαμβάνουν χώρα ε, με νέες προσεγγίσεις, με νέους επεξεργαστές που κατασκευάζονται από αυτούς τους κατασκευαστές δεκτών στο περιβάλλον του Γαλιλαίος για να μπορέσουν να δοκιμάσουν το υλικό τους οι κατασκευαστές και να μπορέσουν να τους διαθέσουν στην αγορά τη στιγμή που το Γαλιλαίος θα μπορεί να λειτουργεί και να παρέχει οι υπηρεσίες. Όσον αφορά την ασφάλεια, που είναι και το θέμα που ενδιαφέρει βασικά την Επιτροπή αυτή, Νομίζω ότι η συνάδελφος ο κ. Άσμπεκ ήδη έδωσε αρκετές πληροφορίες αλλά παρόλα αυτά να επενθυμίσω ένα άλλο σημείο. Το Γαλιλαίος προσφέρει μια υπηρεσία εντελώς ιδιαίτερη. Η υπηρεσία PRS, ε, δηλαδή ε, πρόσβαση δημόσια ρυθμιζόμενη. Η PRS ενσαρκώνει την εξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την δορυφορική πλοήγηση, όπως υπενθυμίζει και ο κανονισμός GNSS του 2013, που είναι ο κανονισμός ε, ο οποίος αναφέρεται και δημιουργεί τα συστήματα τα ευρωπαϊκά δορυφορικής πλοήγης, αυτός ο κανονισμός υπενθυμίζει ότι το PRS αφορά περιορισμένη χρήση, περιορίζεται στους αδειοδοτημένους φορείς ε, που έχουν την άδεια των κυβερνήσεών μας. Επίσης, θα δίνεται και άδεια και στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αυτή η υπηρεσία πιεράς δεν είναι προσβάσιμη παρά μόνο χάρη σε κλειδιά και κάθε κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει κυρίαρχα ποιοι θα είναι οι χρήστες που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κλειδιά, κλειδιά που χρησιμοποιούνται στους δέκτες του PRS ούτως ώστε να αποφεύγεται μια διάδοση ε, διαφόρων συστημάτων, ε, υιοθετούμε αυτό που αποκαλούμε κοινέ προδιαγραφές SNS, Common Minimum Standards, CMS. Ε, είναι στην πράξη της, ε, πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύντομα θα δείτε μια εκδοχή που ελπίζουμε ότι θα είναι η τελική εκδοχή αυτών των κοινών προδιαγραφών. Υπενθυμίζω επίσης ότι σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, πολύ μεγάλης κρίσης, το Συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις σύμφωνα με ένα έγγραφο, μια απόφαση που είναι κοινή δράση και που ε, επικαιροποιήθηκε τον Ιούλιο φέτος. Ε, κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να διορίσει μία αρχή αρμόδια PRS και ήδη έχουμε 14 κράτη-μέλη που καθόρισαν ποια είναι η αρμόδια αρχή PRS που είναι το σημείο επαφής που θα ζητήσει τα κλειδιά πρόσβαση στις υπηρεσίες PRS τα κλειδία πρόσβασης θα ζητηθούν από το κέντρο ασφαλείας και η αρμόδια αρχή PRS θα μπορεί λοιπόν να διανέμει αυτά τα κλειδιά στις ομάδες χρηστών σε κάθε χώρα. Όπως είπε ο Φρανκ Ασμπεκ, το PRS μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, αλλά να επενθυμίσω κάποιους ε, τομείς συμπληρωματικού ε, στους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από τι αστυνομικέ δυνάμεις ε, και από την ακτοφυλακή, από τον έλεγχο των συνόρων, από τα τελωνία, στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, πολιτικής προστασίας για τις περιπτώσεις κρίσης, για κυβερνητικέ μεταφορές, παρακολούθηση επικίνδυνων υλικών, διατήρηση της Ειρήνη, διαφύλαξη Ειρηνή και στην άμυνα. Το PRS έχει χαρακτηριστικά πάρα πολύ ε, ισχυρά έναντι κακών παρεμβολών ε, επιθετικών παρεμβολών και έναντι των καταιγίδων. Ε, λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα σύστημα, το έγνος, το οποίο ήδη λειτουργεί πάρα πολύ καλά και απέδειξε τις δυνατότητες που έχουμε. Το Γαλιλαίος πάντα είναι σε φάση ανάπτυξης και το Γαλιλαίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ε, στο κοινό με ρυθμισμένη πρόσβαση που είναι κλειδί υπηρεσία για την εξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το, ε, το PRS είναι σε κρίσιμο τομέα και θα μπορεί να κινείται συντονισμένη Ευρώπη για την κοινή της ασφάλεια χρησιμοποιώντας το σύστημα PRS. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. Σας ε, ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά. Ο επόμενος ο κύριος Μάουρο Φακίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά παρουσιάστηκαν σχετικά με το Κοπέρνικους. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι ακριβώς λέει το άρθρο 2 του προγράμματος ε, Κοπέρνικος. Δηλαδή το πρόγραμμα Κοπέρνικους ε, είναι ένα πρόγραμμα υπό ε, αστικό έλεγχο και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω γιατί είναι πολύ σημαντικό για την παρουσίασή μου. Βλέπετε λοιπόν εδώ ποιοι είναι κάποιοι από τους στόχους για το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Και βλέπετε ότι πάρα πολλοί εξ αυτών έχουν σχέση με το περιβάλλον, αλλά ε, προστατεύονται επίσης και εγκαταστάσεις ε, και βλέπουμε ότι έχουν και σχέση με την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συνθηκών ασφαλείας. Αυτά έχουν να κάνουν με θέματα ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλιώς αν δεν το φτιάχνατε θα ήμουν αγκασμένος να επισκεφθώ τον ε, οστεοπαθητικό μου. Το Κοπέρνικους ε, προέκυψε με έναν κανονισμό ε, που εκδόθηκε τον Απρίλιο αυτού του έτους και εκδόθηκε και εγκρίθηκε ήδη από την πρώτη ανάγνωση. Άρα δηλαδή είχαμε πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο δραστηριοποιήθηκε στο να γίνουν όλα αυτά δυνατά. Το αποτέλεσμα δεν ήταν τυχαίο, δεν πρόκειψε τυχαία, ήταν το αποτέλεσμα ε, αγαστής συνεργασίας και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα, θα συνεχιστεί και σε αυτό το κοινό κοινοβούλιο. Ο κύριος Πρόντι ήταν ε, ο προηγούμενος συγκητής ε, για αυτόν τον κανονισμό. Έχουμε λοιπόν την ε, λειτουργική φάση του προγράμματος Κοπέρνικους και προβλέπεται ο απαραίτητος προϋπολογισμός για την περίοδο 14 έως 20 και αυτά για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία των δορυφόρων που θα προσφέρουν εικόνες ε, στο σύστημα Κοπέρνικους και επίσης ε, και τα στοιχεία λειτουργίας του να λειτουργούν λοιπόν υπηρεσίες σε σχέση με το Κοπέρνικους. Εδώ στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε περί τίνος πρόκειται στο πρόγραμμα Κοπέρνικους. Πρόκειται για δορυφόρους, τους βλέπετε πάνω δεξιά και πάνω αριστερά. Είναι ειδικοί δορυφόροι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί ε, ειδικά για το Κοπέρνικους. Πρόκειται για τους δορυφόρους που αποκαλούνται Sentinels. Και αυτοί εκτελούν αποστολές είτε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε αλλού. Υπηρεσίες λοιπόν. Οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή ομαδοποιούνται σε έξι τομείς τους οποίους ε, τρεις εξ αυτών ε, καλύπτουν τις ε, βασικές φυσικές παραμάτρους της γης, δηλαδή τη γη, την ατμόσφαιρα και τη θάλασσα. Άλλοι τρεις ε, καλύπτουν ε, οριζόντιες ανάγκες, έκτακτες ανάγκες, ε, κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια. Και όσον αφορά την ασφάλεια θα επανέλθω. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα τύχει διαχείρισης αποκεντρωμένης. Και πάμε στην επόμενη διαφάνεια και βλέπουμε όλους τους φορείς που θα εμπλακούν ε, στην ε, διαχείριση του Κοπέρνικους. Έχουμε λοιπόν τους δορυφόρους και θα συνεργαστούμε με την ε, Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Επίσης θα συνεργαστούμε με τους περισσότερους διαστημικούς φορείς που υπάρχουν στην Ευρώπη για να έχουμε δεδομένα. Και όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βασιστούμε στους σημαντικότερους οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Για τη γη βασιζόμαστε ε, ε, στον οργανισμό που υπάρχει στην Κοπενχάγη. Τώρα, για την κλιματική αλλαγή ε, θα βασιστούμε στον οργανισμό που υπάρχει στο Reading, στο Ηνωμένο Βασιλείο και για το, το, τμήμα της θάλασσας στον αντίστοιχο φορέα που υπάρχει στη Γαλλία. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, θα συνεργαστούμε με τη Frontex. Όσον αφορά την επιτήρηση των συνόρων με την ΕΜΣΑ για τη θαλάσσια επιτήρηση και ο Φρανκ Ασπέκ αναφέρθηκε και στο ε, δορυφορικό κέντρο, κυρίως όσον αφορά τις δράσεις του, τις εξωτερικές του δράσεις. Τώρα θα μπω με λεπτομέρειες σε, σε θέματα ασφάλειας πιο κοντά σε αυτά που βρισκόμαστε σήμερα. Ο κανονισμός Κοπέρνικους αναφέρει ότι η υπηρεσία ασφάλειας ε, που θα είναι μία από τις έξι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι να προσφέρει πληροφορίες για τις απειλές ασφάλειας στην Ευρώπη ε, συμπεριλαμβανομένης βελτίωσης της πρόληψης κρίσεων, της ε, προετοιμασίας κυρίως ε, για την επιτήρηση στα σύνορα, στη θάλασσα αλλά και στις εξωτερικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή πρόκειται για υποστήριξη αυτών των τριών πολιτικών. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάποια παραδείγματα εικόνων που δείχνουν με πολύ απλό τρόπο το τι μπορούμε να δούμε ε, κατά την επιτήρηση των συνόρων της θάλασσας και των εξωτερικών δράσεων. Και αυτά ε, τα στοιχεία προσφέρονται στους εμπειρογνώμονες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την πολιτική τους και για εσωτερική χρήση. Αναφέρθηκα λοιπόν σε τρεις τομείς, στην επιτήρηση των συνόρων, αυτό είναι ο πρώτος τομέας. Και αυτός είναι ένα εργαλείο για να στηρίξουμε τη Eurosur. Και γι' αυτό ε, διαπραγματευόμεθα με τη Frontex ε, έτσι ώστε ε, να εκχωρήσουν αυτό το εργαλείο, όμως η Frontex ε, δεν θα λειτουργεί μόνη της σε συνεργασία με την ΕΜΣΑ και με το Δορυφορικό Κέντρο. Με την ΕΜΣΑ για τα σύνορα στη θάλασσα και το Δορυφορικό Κέντρο για την επιτήρηση των σύνορων, των χερσαίων σύνορων. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο σε αυτά που ήδη κάνει η Frontex ε, στον τομέα της επιτήρησης των συνόρων με την έννοια ότι υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερη εποπτεία σε αυτόν τον τομέα. Μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις όπως η παράνομη μετανάστευση. Εξετάζοντας όλα αυτά προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος και επίσης ε, αναζητάμε και αποτελέσματα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο project αλλά όλα αυτά θα μπορούν αργότερα να ενταχθούν και ε, στην πράξη. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει είναι η θαλάσσια επιτήρηση. Πρόκειται εδώ για μια ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση του ε, κοινού περιβάλλοντος ενημέρωσης αλλά και πάλι στηρίζουμε την επιτήρηση των συνόρων ε, στη θάλασσα, ε, χερσαία επιτήρηση και πάρα πολλά παρεμφερή. Αυτές δηλαδή είναι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο ΕΜΣΑ και γι' αυτό η ΕΜΣΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για όλες αυτές τις δράσεις. Και πάλι, όπως και με τη Frontex, διαπραγματευόμαστε μία συμφωνία με την ΕΜΣΑ. Το τρίτο που μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ περιλαμβάνεται η αντίδραση στις κρίσεις, η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, η ενίσχυση της δημοκρατίας, ενευτικών διαδικασιών και το καθεξής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσφέρουμε στήριξη της ευρωπαϊκής πολιτικής στις εξωτερικές της δράσεις. Και πάλι προσφέρουμε επιπρόσθετες πληροφορίες ε, για να στηρίξουμε όλα αυτά που προανέφερα. Όπως σας είπα λοιπόν, όσον αφορά το πρόγραμμα εφαρμογής, ε, έχουμε τρεις τομείς, επιτήρηση των συνόρων, θαλάσσια επιτήρηση, και για τις εξωτερικές δράσεις. Εκεί βεβαίως και προσφέγουμε στην ε, διακυβέρνηση του συστήματος, αλλά το δορυφορικό κέντρο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Όταν μιλάμε για εκχώρηση, κατ' ουσίαν αυτές, αυτοί οι οργανισμοί θα ασχοληθούν με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, αλλά τα χρήματα θα παραμείνουν απλά σε αυτά αυτούς τους οργανισμούς απλά θα δοθούν για να συναυτούν τα απαραίτητα συμβόλαια και να προσφερθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες. Όσον αφορά την πολιτική των δεδομένων, αυτή αφορά το πρόγραμμα Κοπέρνικους και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί γίνεται. Γιατί ο πρώτος λόγος είναι ότι τα περισσότερα στοιχεία ε, που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος Κοπέρνικου δεν είναι εμπέστητα. Έτσι λοιπόν, το να προσφέρουν τα στοιχεία δωρεάν υπάρχει η δυνατότητα να συσταθεί και μια συγκεκριμένη αγορά γιατί μερικές φορές ε, υπάρχουν στη μία μπλοκαρίσματος για να δημιουργηθεί μια κάθετη αγορά ε, και αυτό οφείλεται κυρίως στην τιμή. Εδώ πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Και γι' αυτό υπάρχει και ένας κανονισμός που αναφέρεται σε αυτή την πολιτική δεδομένων. Όμως σε αυτή την πολιτική πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα σε διάφορα στοιχεία, δηλαδή τα δεδομένα των ειδικών δορυφόρων ε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται για το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Έχουμε τα προϊόντα του Κοπέρνικου που είναι δωρεάν και ελεύθερα με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Έχουμε και ε, κάποιες ειδικέ αποστολές. Εκεί τα δεδομένα εξαρτώνται από τους παρόχους γιατί υπάρχουν κάποιες ε, προϋποθέσεις αντιοδότησης που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Παρότι λοιπόν ε, όλα αυτά βλέπονται δωρεάν υπάρχουν και κάποιες ε, προϋποθέσεις ασφάλειας. Και αυτός είναι ο λόγος γιατί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις έκτακτες ανάγκες εκτός Ευρώπης για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν όλα αυτά είναι ευαίσθητα και αυτά πρέπει να εξεταστούν με μεγαλύτερη ευαισθησία ε, σε σχέση με την εξωτερική δράση. Ένα λοιπόν από τα άρθρα του κανονισμού, το άρθρο 25, προβλέπει την αξιολόγηση του ε, πλαισίου του Κοπέρνικους και αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια μελέτη τα ε, αποτελέσματα προβλέπονται για το 2015. Αυτά είχα να σας πω. Ε, μία μόνο διαφάνεια θέλω να σας δείξω ακόμα που αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους για το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Το κόστος λοιπόν, είδαμε τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα Κοπέρνικους, αλλά στη τελική ανάλυση το διάστημα είναι κάτι δαπανηρό γιατί όταν μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια ή 7 δισεκατομμύρια για το Γαλιλαίος, αν δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στους διάφορους τομείς και υπολογίσουμε το κόστος, θα διαπιστώσουμε ότι το κόστος είναι περίπου ένα ευρώ ανά Ευρωπαίο πολίτη για να επιτύχουμε όλα αυτά που σας προανέφερα και πάνω από τα οικονομικά ωφέλη που εκτιμώνται σε πολλά δισεκατομμύρια θα δημιουργηθούν 40 ε, μέχρι 50.000 θέσεις εργασίας, απασχόλησης. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε βέβαια να τα αναλύσουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτά είναι καθαρά υποκειμενικά. Γιατί αν δούμε τις επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, ζωές που μπορούν να σωθούν από μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ε, μετρηθούν ποσοτικά. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει την αξία της ζωής ενός ανθρώπου που ε, μπορούμε να σώσουμε με μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ κύριε Φακίνη. Ξεκινάμε τη συζήτηση κ. Ντονζόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Έγιναν πολλές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων για την διαστημική πολιτική και ποια είναι η διάσταση ασφάλειας και άμυνας του διαστήματος. Η ομάδα μου και εγώ δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτή την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική και τη συνιστόσα της στην αμυντική. Πάντα ζητούσαμε κάτι τέτοιο να γίνει και για τα διάφορα προγράμματα. Λυπούμε που επανέρχομαι πολύ συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα της εκτόξευσης δορυφόρων το καλοκαίρι αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα από αυτά που μας είπατε. Να εκφράζω την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά για τις επόμενες εκτοξεύσεις, μπορούμε να ελπίζουμε, και τελικά ακόμα και αν δεν φτάσουμε στην τροχιά, την αρχικά προβλεπόμενη, να πλησιάσουμε. Θα ήθελα να μας υπενθυμίσετε όμως κάτι, διότι έγινε Επιτροπή Έρευνας. Ποια δυσλειτουργία απεκαλύφθη από αυτό το πρόβλημα. Διερωτώ με πάντα εγώ, πολιτικός πώς, όσον αφορά την επιλογή των πυράβλων Σογιούς, θα πρέπει να το πανεξετάσουμε και αυτό, διότι το Κοπέρνικος, μάλλον το Γαλιλαίο, συγγνώμη λέει ο μιλητής, μας πουλήθηκε κυριολεκτικά πουλήθηκε. Και εμείς οι πολιτικοί πουλάμε το Κοπέρνικους, το Γαλιλαίος, συγγνώμη λέω το πουλάμε σαν ένα μέσο βασικό εργαλείο στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πάρα πολύ ακριβό πρόγραμμα που δημιούργησε προβλήματα σε κάποια κάτι μέλη για τη χρηματοδότησή του και κάθε φορά αυτοί που υπερασπίζονται το πρόγραμμα, μεταξύ αυτών και εγώ, βγήκαμε ε, στην πρώτη γραμμή του υπερασπιστούμε και είπαμε ότι είναι απαραίτητο εργαλείο για την ευρωπαϊκή ε, στρατηγική, για την ανεξαρτησία της. Και ε, υπάρχουν διαμαρτυρίες διότι αναμειγνύουμε ξένες δυνάμεις. Ε, και δημιουργούμε συμμαχίες που ελπίζω στην Κυριακή Συμμαχία που είναι όμως πολύ ενοχλητική ε, λόγω της κρίσεως που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αναφέρθηκα στο ιστορικό λοιπόν αυτής της συνεργασίας με το Ισογιούς και θα ήθελα να γνωρίζω ποιες είναι οι αναμενόμενες εξελίξεις όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Thank you, Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ενημερώσεις που μας έκαναν. Διαπιστώνω εξέλιξη. Θυμάμαι ότι υπήρχε μεγάλος δισταγμός να δεχτεί η Υποπιτροπή ότι είναι ζήτημα το Γαλιλαίος. Ότι το πρόγραμμα απαιτούσε μία σφαιρική προσέγγιση από την Ένωση και χρηματοδοτικά. Να υπάρχει κοινή χρηματοδότηση. Και έπαιξε το ρόλο του το Κοινοβούλιο στο να περάσει η κοινή χρηματοδότηση. Γι' αυτό και τότε τα προγράμματα ήταν απλώς πολιτικά, δεν εκάλυπταν το στρατιωτικό τομέα. Ήταν προφανές ευθύς εξ αρχής όμως ότι σχετιζόταν το στρατιωτικό τομέα. Ότι σχετιζόταν με τη στατική μας αυτονομία, με την ασφάλεια και την άμυνά μας. Και είναι αρκετά θετικό το, από αυτά που ακούσαμε το ότι τώρα υποτίθεται πλέον ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε από τη μία πλευρά δηλαδή την πολιτική προστασία, την άμυνα τα οποία είναι αλληλένδετα. Και πρέπει να πω ότι ο ρόλος των προγραμμάτων, των διαστημικών και των σχετικών συναφών εφαρμογών όπως δορυφορική πλοήγηση, το έγνος είναι σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά και για την εξωτερική πολιτική. Υπενθυμίζω τη σημασία της δορυφορικής φωτογράφησης για την ειρηνευτική ε, διαδικασία στο Χάτσε όταν είχαμε όταν ήταν τους τυφώνες και στην Ινδονησία οι τοπικές αρχές μπορούσαν να βρουν συγκεκριμένα ε, τις περιοχές που είχαν καταρρεύσει τα σπίτια και μπόρεσαν οι άνθρωποι να βοηθηθούν και να βρουν τις ε, ιδιοκτησίες τους και να μην περιπλακεί περαιτέρω η κατάσταση η κυρινευτική διαδικασία. Υπάρχει η ειρήνη στο Άτσε, έπαιξε το ρόλο της έπαιξε το ρόλο της και το κοινοβούλιο. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, και είναι σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Ντανζάν για την εξάρτησή μας από άλλες δυνάμεις. Κυρίως όταν οι άλλες δυνάμεις αυτές βλέπουμε ότι δεν είναι πραγματικά αξιόπιστες, αξιόπιστοι εταίροι. Πρόσφατα είχαμε σειρά πτήσεων υπερπτήσεων από ρωσικά αεροσκάφη, στρατιωτικά αεροσκάφη, πάνω από τον εναέριό μας, από την επικράτειά μας, το δικό μας εναέριο χώρο. Και πέρσι αυξήθηκε το φαινόμενο των παραβιάσεων του εναερίου χώρου. Αυξήθηκαν οι παραβιάσεις και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους και για την πολιτική αεροπορία. Έχουν συγκεκριμένη περίπτωση όπου χρειάζονται τα συστήματα. Να εντοπίζουμε και να προστατεύουμε, να αναχαιτίζουμε και να προστατεύουν την επικράτειά μας. Αναφέρθηκε η έκθεση των δυνάμεών μας και των αποστολών μας ε, στο εξωτερικό. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα συστήματα γι' αυτό. Η θαλάσσια υποπτία. Όταν έκανα την έκθεση για την ε, θαλάσσια διάσταση, το διαπίστωσα αυτό. Αναφέρθηκατε στην σημασία που έχει η ΕΜΣΑ. Η ΕΜΣΑ έκανε πολύ σημαντικά πράγματα για την προστασία μας, για την άμυνά μας. Η ΕΜΣΑ δεν είχε εντολή για κάτι τέτοιο όμως και βλέπω ότι τώρα πια άλλαξαν τα πράγματα. Όχι εντολή, αλλά η προσέγγιση είναι κάπως διαφορετική. Ερώτηση. Οι, οι κυβερνήσεις μας αναγνωρίζουν τι διακυβεύεται. Κυρίως αυτά που ανέφερε ο κ. Χάσμπεκ. Αντιμετωπίζουμε πραγματικές απειλές. Κάθε είδους και κυβερνοαπειλές. που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τον τρόπο ζωής μας, τις κρίσιμες υποδομές μας, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τα κράτη-μέλη το καταλαβαίνουν. Βλέπω κάποια κράτη-μέλη, κυρίως ένα κράτο, τη Βρετανία, δεν θα το αποκρύψω, να θέτουν εμπόδια. Σε αυτά πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να παράσχει τα προγράμματα αυτά που επιτυγχάνονται μέσω ευρωπαϊκής σύμπραξης. Και βλέποντας τεράστιες οικονομικές περικοπές που γίνονται παντού, σε όλες τις χώρες. Εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κυβερνήσεις μας καταλαβαίνουν τι διακυβεύεται. Η ερώτησή μου είναι αυτή. Αισθάνεστε ότι οι κυβερνήσεις μας το καταλαβαίνουν αυτό. Τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων στον τομέα αυτό, στα προγράμματα αυτά. Μας παρουσιάσατε. Thank you, madam. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Κάμπελ Μπάνεμαν, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαν οι καλεσμένοι μας, αλλά διερωτώ με το κόστος του Γαλιλαίου. 20 δις ευρώ για 20 χρόνια εκτιμάται. Και το μεγαλύτερο κόστος είναι για την ανάπτυξη και όχι για την λειτουργία του. Οι δορυφόροι είτε θα μπουν όμως υπάρχει κίνδυνος σε λάθος τροχιά είτε από ό,τι με έχουν ενημερώσει δεν θα μπορούν να μετακινηθούν στη σωστή τροχιά. Άρα θα είναι άχρηστοι για το σκοπό που θα έχουν εκτοξευτεί. Διερωτώμε λοιπόν το κόστος αυτού του προγράμματος. Πώς ε, αιτιολογείται γιατί δεν χρησιμοποιούμε το σύστημα απλοηγήσης ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί δαπανάμε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, όπως είπε και η κυρία Γκόμες. Εμένα με απασχολεί ας πούμε το ότι η Wikileaks ε, έχει παραθέσει κάτι από μια γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει αυτούς τους δορυφόρους που λέει ότι κατά την άποψή τους το πρόγραμμα Galileo είναι μια νόητη ιδέα που κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τα γαλλικά συμφέροντα και σπαταλά τα χρήματα του φορολογούμενου. Εντάξει, όχι ότι, ό,τι λέει το Wikileaks είναι Ευαγγέλιο, αλλά μήπως το λέει σωστά. Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας επισημάνω το θέμα της ασφάλειας. Για μένα λοιπόν είναι καθοριστική σημασίας ότι θα πρέπει να επισημάνουμε με σαφήνεια όσον αφορά το κόστος πάντα, ποιο είναι το στοιχείο της ασφάλειας αυτού του δορυφορικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και όλες οι απειλές ε, να αποφευθούν. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι εγώ συμφωνώ το πρόγραμμα Κοπέρνικους πρέπει να ε, κατασκευαστεί, να εφαρμοστεί. Ό,τι είδαμε σήμερα πρέπει να προετοιμαστεί αξιόπιστα έχοντας πάντα κατά νου την ασφάλεια. Επίσης έχοντας κατά νου όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την οικονομική ανάπτυξη και για την ασφάλεια. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι ο λόγος που παίρνω το λόγο είναι ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες για θέματα συνεργασίας μέσα σε αυτό το σύστημα και υπάρχουν και κάποιες υπόνοιες ε, για ε, σκόπιμες ε, παρεμβολές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μιλτές, αλλά την πρώτη ερώτηση θα ήθελα να την απευθύνω προς τον κύριο Πολ Φλαμό. Δηλαδή, το σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί πλήρως και το οποίο βασίζεται στο αμερικανικό σύστημα GPS αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο βελτιώνεται συνεχώς, δηλαδή το πρόγραμμα Γαλιλαίος ε, είναι συμβατό με το σύστημα GPS. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζω είναι το εξής κατά πόσον ενδεχομένως πρόκειται να αντικαταστήσουμε το σύστημα έγνος από το σύστημα Γαλιλαίος. Και να κάνω και μία πολιτική φύσεως ε, δήλωση μετά την παρέμβαση του κ. Νταζόν με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κατασκευή του συστήματος Γαλιλαίος ο λόγος που κατασκευάστηκε αυτό το σύστημα είναι κυρίως για να είμαστε ανεξάρτητοι. Όμως βλέπουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι θέλαμε να ανεξαρτητοποιηθούμε από ένα πολύ μεγάλο εταίρο από τις Ηνωμένε Πολιτείες όμως με τον εταίρο μας αυτό έχουμε πολλές συμφωνίες σε άλλους σημαντικούς τομείς τομείς ε, οι οποίοι και αυτοί πάλι έχουν άμεση σχέση με τα συστήματα και τα προγράμματα που συζητάμε. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη, το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών φιλοδοξιών είναι το εξής. Έχουμε συστήσει σχέσεις ε, με έναν εταίρο, ο οποίος αποδεικνύεται όχι μόνο απρόβλεπτος, Δηλαδή δεν είναι αξιόπιστος ο εταίρος μας και το ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στις ΗΠΑ αυτό είναι το λιγότερο μπορούμε να πούμε. Έχουμε να κάνουμε με έναν εταίρο ο οποίος παραβιάζει τον ενέριο χώρο μας ε, και αυτό μάλιστα σοβαρά σε πάρα πολλούς ε, σε πάρα πολλές τοποθεσίες μέσα από ε, στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί κίνδυνο για τους ε, υπηκόους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας εταίρος ε, ο οποίος είναι, επιτίθεται σε αυτούς που έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με μας. Επίσης, ο εταίρος αυτός αποτελεί κίνδυνο για πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και υπάρχουν ανησυχίες που εκφράζονται σε κάθε λομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν έχω μία ερώτηση να απευθύνω προς όλους σας. Γνωρίζω ότι είσαστε εμπειρογνώμονες σε αυτό τον τομέα, αλλά θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι αναθεωρημένη ανάλυση του συνόλου του πολιτικού συστήματος έχοντας κατά κύριο λόγο κατά νου αυτή τη συνεργασία που σας ανέφερα. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα να κάνω μία άτυπη ερώτηση προς την Επιτροπή και προς ε, την ύπατη εκπρόσωπο. Η ερώτηση μου αφορά το κόστος. Το κόστος ε, ενός τέτοιου εγχειρήματο. Όχι μόνο τα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί στο σύστημα γιατί κανείς που είναι λογικός δεν θα ε, παρατηθεί ενός προγράμματος το οποίο μας έχει κοστίσει όχι μόνο τόσες πολλές προσπάθειες αλλά και όλους αυτούς και τους οργανισμούς που λειτουργούν αλλά μας έχει επίση κοστίσει και χρήματα γι' αυτό η ερώτησή μου είναι η εξής είναι μία ερώτηση προς τον κύριο Ντανζό. Δηλαδή αυτό το σύστημα το οποίο τώρα χρησιμοποιείται στη Γαλλική Γουινέα αυτό το σύστημα σημαίνει ότι θα έχουμε την εκτόξευση νέων δορυφόρων. Δεν θα φτάσουμε ε, στους Σόγιους πριν εκτοξευτούν οι Αριάν και αυτό δεν είναι λόγος για να πάψει να ισχύει η συμφωνία. Oh. Now I would like to... Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ να απαντήσουν ερωτήσεις. Α, ο κύριος Ντανζόν παρακαλώ όμως πρώτος. Ζήτω συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί μου θέσατε ερώτηση. Δεν κατάλαβα, είμαι Γάλλος. Δεν διευθύνω το κουρού, τη βάση του κουρού, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Η εθνικότητά μου δεν έχει σχέση με την ερώτησή μου όσον αφορά το Γαλιλαίος και τους πυράβλους για την εκτόξευση δορυφόρων. Ευχαριστώ. Mr. first and then... κύριε Άσπεκ πρώτος και μετά ο κύριος Φλαμάου, μετά ο κύριος Φακίνη να απαντήσετε τις ερωτήσεις παρακαλώ. Εντάξει σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για τα ευγενικά σχόλια και αναφέρομαι ιδιαίτερα στα σχόλια που έγιναν από την κυρία Γκόμες για τον ρόλο που διαδραμάτισε το δορυφορικό κέντρο κατά το παρελθόν. Τώρα, θα προσπαθήσω πρώτα να απαντήσω το ερώτημα για την συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της ασφάλειας για τα διαστημικά θέματα. Συμφωνώ μαζί σας ότι, πώς να το πω, το επίπεδο ευαισθητοποίησης για τη σπουδαιότητα των θεμάτων ασφάλειας στα διαστημικά θέματα διαφέρει πάρα πολύ από κράτος σε κράτος και φυσικά μεταξύ των κρατών μελών έχουμε και εκείνα που εμπλέκονται πιο πολύ στα διαστημικά θέματα και εκείνων που εμπλέκονται λιγότερο. Όμως πιστεύω ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι τελικά να αυξήσουμε το επίπεδο ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης όλων των κρατών. Το ότι όλοι εξαρτόμαστε από υπηρεσίες διαστημικές σήμερα και πρέπει φυσικά να είναι για αυτόν τον λόγο προς το συμφέρον όλων να διασφαλίζουμε ότι τα διαστημικά συστήματα δορυφορικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε λειτουργούν από επιμέρους κράτη-μέλη είτε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά οι πτυχές της ασφάλειας διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει πάντα να το θυμόμαστε αυτό. Επίσης, η συνολική η σύνολη κατάσταση όπως έχει για τα διαστημικά θέματα της διαστημικής μπορεί να δυσχερανθεί λόγω διαφορετικών λόγων στο μέλλον περισσότερο. Και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και εγχειρήματα που βρίσκονται υπό εξέλιξη Σίγουρα καλωσορίζουμε τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ σήμερα, διότι συνεισφέρει να αυξηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίηση σίγουρα, αλλά καλωσορίζουμε και οποιαδήποτε συζήτηση με τη συμμετοχή των κρατών μελών για την ανάγκη να προχωρήσουμε και να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Και θα υπάρξει και συζήτηση στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας κατά το δεύτερο ε, ήμιση του Νοεμβρίου και θέματα διαστημικής και ασφάλειας στα διαστημικά θα καλυφθούν και εκεί. Αυτά για αυτό το ζήτημα. Φοβούμαι ότι δεν είμαι σε θέση να απαντήσω το ερώτημα όσον αφορά την εντολή ένσας. Ωστόσο όμως φυσικά το συνολικό ζήτημα της ε, ναυτιλιακής ε, παρακολούθησης και εποπτείας και της μεγάλης σημασίας του όλο και περισσότερο μας αναφέρεται και από εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε διαλόγους ε, για διαφορετικά θέματα και σε διαφορετικά επίπεδα με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και βλέπει κανείς από όλα αυτά ότι η χρήση του διαστήματος για την ναυτική, ναυτιλιακή εποπτεία και η αύξηση της συνειδητοποίησης και της ευαισθητοποίησης της σπουδαιότητάς τους είναι πολύ σημαντικό θέμα και όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα αποκτά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα, το θέμα της χρήσης, πώς να το αποκαλέσω, το σύστημα Γαλιλαίος έναντι του GPS και δεν κάνω εδώ λόγο για θέματα κόστους-οφέλους γιατί αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχει πολύ μεγαλύτερα, ε, μεγαλύτερες γνώ, περισσότερες γνώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί από αυτού, αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι πριν από 10 χρόνια περίπου υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την πλευρά των ΗΠΑ, της ΗΠΑ σε σχέση με το εγχείρημα αυτό, το σχέδιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση αυτή άλλαξε άρδιν δραματικά και στις ε, τακτικές μας επαφές και ανταλλαγές απόψεων με τη ΣΥΠΑ οι ΙΠΑ εκφράζουν την ικανοποίησή τους ότι μια ομάδα κρατών όπως ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσουν τώρα αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύστημα το οποίο συμπληρωματικά και παραπληρωματικά θα λειτουργεί σε σχέση με το GPS, το σύστημα εντοπισμού στίγματος από πλευρά των ΗΠΑ. Ενδιαφέρονται οι ΗΠΑ να συνεργάζονται στενά και να συνεργαστούν στενά με, τις, ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πεδίο. Το θέμα της συμπληρωματικότητας, ε, ε, παραπληρωματικότητας είναι σημαντικό. Φυσικά λόγω της αυξημένης εξάρτησης της ανθρώπινης ζωής των ανθρώπων από την δορυφορική ναυτιλία για παράδειγμα. Είχαμε περιπτώσεις, είχαμε και μια περίπτωση όπου απέτυχε το ρωσικό σύστημα εντοπισμού για μια μέρα για να παράσχει τέτοιου είδους στοιχεία και ε, πληροφορίες στίγματος ε, και εντοπισμού. Μπορείτε να φανταστείτε που οδηγεί κάτι τέτοιο ή που θα οδηγούσε αν αποτύχανε να λειτουργήσει το GPS και ε, έπαβε να λειτουργεί όλοι θα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι να είχαν ένα σύστημα αναδίπλωσης, σύστημα εφεδρικό, αμοιβό σύστημα χρήσης. Και εδώ θα πρέπει να το δούμε αυτό. Μήπως θα υπάρξουν κάποιοι λόγοι που θα, αναγκού, αν, θα καθιστούσαν αναγκαίο για τις να αλλάξουν κάποια στοιχεία στα επίπεδα και στη χρήση του GPS σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί να αφαιθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία δορυφορικής ναυτιλίας και εντοπισμού στίγματος. Είναι κρίσιμη σημασία και θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν για τη διασφάλισή τους οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά για να απαντήσω σε σχέση με αυτό το ζήτημα απόλυτα ανεξάρτητα από την οικονομική συνιστόσα παράμετρο αυτού του θέματος είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική επένδυση την οποία ακολουθεί και καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα θέματα. Μπορώ να δώσω νομίζω τώρα τη σκητάλη σε άλλον. Ευχαριστώ. Κύριος Φλαμό τώρα παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Γκόμες αφορούσε τις πτυχές ασφάλειας και αν τα κράτη-μέλη έχουν επίγνωση σημασίας που έχει ασφάλεια. Απάντηση είναι απλούστατη ναι. Να σε εξηγήσω γιατί όσον αφορά το Γαλιλαίος αυτό υλοποιείται και φαίνεται έχουμε πολλά μέσα, πολλά εργαλεία που υπάρχουν και που 100% εμπλέκουν τα κράτη-μέλη στη σύλληψη του συστήματος Γαλιλαίος και στην επαλήθευση του κατά πόσο είναι ασφαλές. Έχουμε μία επιτροπή η οποία επιβάλλει περιορισμούς και όρους συνδέονται με την ασφάλεια στο σύστημα Γαλιλαίος. Διότι τα κράτη-μέλη έχουν την εμπειρία επί του θέματος και συμβάλλουν τι ο τρόπος λέγοντας ποιες απαιτήσει συγκεκριμένες έχουν για να συμμορφωθεί το Γαλιλαίος. Όταν θα ολοποιηθεί το σύστημα, πριν γίνει επιχειρησιακό, τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν στην, ε, στην έγκρισή τους όσον αφορά την ασφάλεια. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών, οι οποίοι θα δώσουν την άδειά τους ή την άρνησή τους ε, για την τοποθέτηση ενό δορυφόρου ή τη δημιουργία κέντρου ελέγχου. Έχουμε την Επιτροπή ε, Διαπίστωση Εξακρίβωσης Ασφαλείας, Έγκρισης Ασφαλείας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών. Μετέχουμε κοινή δράση που ε, συνεπάγεται εμπλοκή και του Συμβουλίου και έχουμε διάφορα μέσα, ε, έχουμε τα κέντρα ασφαλείας, έχουμε ένα διπλό κέντρο ασφαλείας στην Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, όσον αφορά το επίμαχο θέμα της ύπαρξης ή του λόγου ύπαρξης ή μη του Γαλιλαίος, από το 2004 πράγματι έχουμε συμφωνία με τους Αμερικανούς και αν έχουμε αυτή τη συμφωνία με τους Αμερικανούς είναι διότι αυτοί οι ίδιοι αναγνωρίζουν το συμφέρον να υπάρχει και άλλο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης πέραν του GPS. Να θυμηθούμε ότι το σύστημα παραμένει εύθραυστο, είναι εύθραυστα σημεία, δύσκολο να δημιουργηθούν. 20 χρόνια χρειάστηκαν οι ΙΠΑ για να δημιουργήσουν το GPS. Οι Ρώσοι ήδη πάνω από 120 δορυφόρους γκλονάς εκτόξευσαν πριν να φτάσουν κάτι που να λειτουργεί λίγο πολύ παραμένει μια υποδομή χρήσιμη σε ενιαία σε μοναδική βάση αν έχουμε μια τέτοια υποδομή θα ήταν κάτι συνείδητο και επικίνδυνο. 7% του ΑΕΠ των συγχρόνων οικονομιών δράζεται επί της χρήσης των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης. Και κάτι τελευταίο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί πλήρως το σύστημα Γαλιλαίος, διότι η βιομηχανία της, του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχει πλήρως στην υλοποίηση του Γαλιλαίου. Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση, για την αποστολή σημάτων στο Γαλιλαίο παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει και μια μονάδα παραγωγής μηχανημάτων στο Στάνουικ. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θέτησαν κανονισμό ο οποίος στηρίζει και ε, δημιουργεί και υλοποιεί το σύστημα Γαλιλαίος όσον αφορά το πιο συγκεκριμένο ερώτημα του κυρίου Ντανζάν που αφορούσε τις εκτοξεύσεις. Καταρχάς πρέπει να γνωρίζετε ότι η υπηρεσία εκτοξεύσεων είναι κάτι παρακινδυνευμένο. Θα είδατε εικόνες αρκετά θεματικές την περασμένη εβδομάδα της εκτόξευσης της ΕΠΑ από την Orbital Science, από την εταιρεία Orbital Science που πύραυλωσε εξεράγει λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση και η Virgin Galactic και άλλη εταιρεία που δημιουργεί το Spaceship 2 αντιμετώπισε προβλήματα. Η εκτόξευση δορυφόρων, η εκτόξευση αντικειμένων στο διάστημα πάντα ήταν κάτι επικίνδυνο και το επίπεδο αξιοπιστία των καλύτερων πυράβλων στον κόσμο, που είναι η Σογιούς και η Αριάν 5, είναι της τάξης 97%. Πάντα υπάρχει ένα 3%, τρεις εκτοξεύσεις από τις 100 που οδηγούν σε αποτυχία. Η εκτόξευση έλαβε χώρα περίπου 20 Αυγούστου από τη Γαλλική Γουιάννα με πύραυλο Σογιούς. Ο Σογιούς έθεσε τους δύο δορυφόρους Γαλιλαίος σε κακή τροχιά. Αμέσως μετά από αυτό η εταιρεία Ariane Spass που είναι υπεύθυνη για τη σύμβαση και για τις εκτοξεύσεις αμέσως ε, ε, δημιούργησε μια επιτροπή έρευνας. Στην επιτροπή έρευνας έχουμε τουλάχιστον 10 μέλη στην επιτροπή έρευνας μεταξύ των οποίων μεγάλο ειδικό του διαστήματος ο κ. Πίτερ Ντιμπόκ, ε, που ήταν Γενικό Επιθεωρητή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο, συνοδευόμενο από μεγάλου ειδήμονε αρκετών κρατών μελών, ε, Γάλλου, ε, Βρετανού, Ιταλού, Γερμανού, ειδικού που πήγαν εκεί και αυτά τα μέλη έκαναν μία έρευνα. Και ο πελάτη εκπροσωπεί και εγώ προσωπικά συμμετείχα σε αυτή την ερευνητική επιτροπή σαν μέλος. Ε, ε, έγιναν πάρα πολλές συνεδριάσεις και στην έδρα της Αριάνες Πας και στη Μόσχα, στα γραφεία της Γκλαφς Κόσμος για να αναλύσουμε όλα τα στοιχεία που διαθέταμε σχετικά με αυτό το γεγονός. Ε, ε, είδαμε στοιχεία τηλεμετρικά, εξετάσαμε πληροφορίες αυτού του τύπου από τον ίδιο τον ε, πύραυλο που μας στείλανε Είδαμε διάφορα τα σχήματα, τα σχέδια του συστήματος και εξετάσαμε διάφορα ενδεχόμενα, κάναμε προσωμιώσεις κλπ. Ούτως ώστε τελικά να βρούμε ποιο ήταν το αίτιο του προβλήματος που αντιμετωπίζαμε. Προφανώς είμαστε πιο ευφυείς μετά από το γεγονός και το πρόβλημα καταλαβαίνοντας τι συνέβη. Το πρόβλημα είναι απλούστατο, επρόκειτο περί δύο σωλήνων που συνδυόταν ο ένας με τον άλλον, ενώ δεν έπρεπε να είναι συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον. Και για λόγους ε, ε, θερμικών προβλημάτων, το υδραζίν, ένα προϊόν που χρησιμοποιείται, ε, πάγωσε ε, για κάποιο χρονικό διάστημα και αυτό το παγωμένο υλικό μετά από κάποιο χρόνο οδήγησε στο να τεθούν οι δορυφόροι σε λάθος ε, ε, τοποθέτηση, σε λάθος τροχιά. Μπορώ να σα δώσω και άλλε λεπτομέρειε. Αν κάποιοι ενδιαφερόσαστε με ένα καφεδάκι, σα εξηγώ τι λεπτομέρειε μετά. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν λοιπόν στην ερευνητική αυτή επιτροπή, την Επιτροπή Έρευνα, ξέρουν ακριβώ ποια είναι η προέλευση του προβλήματο. Είναι ένα πρόβλημα τεχνικό, όσον αφορά το σχεδιασμό η εταιρεία εκτόξευσης για Πας ε, ανέλαβε κάποιες δράσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα και έτσι μπορούν ξανά να λειτουργήσουν σωστά οι πύραυλοι Σογιούς. Την περασμένη εβδομάδα οι Ρώσοι που χρησιμοποίησαν πύραυλο Σογιούς ακριβώς τον ίδιο με αυτόν που χρησιμοποίησαμε εμείς έκαναν εκτόξευση ένα κυβερνητικό δορυφόρο, τον μεριδιάν εκτόξευσαν και η εκτόξευση λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Αυτό το μήνα οι Ρώσοι εκ νέου χρησιμοποίησαν τον πύραυλο Σογιούς με τον ίδιο με τρόπο όπως και εμείς για να εκτοξεύσουν δύο ε, δορυφόρους Και το Δεκέμβριο ο πύραυλος Σογιούς θα εκτοξευτεί εκ νέου από τη γαλλική βάση στη γαλλική Γουιάννα, στο Κουρού και θα μεταφέρει εμπορικό φορέα τον E3B η SS Άστρα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος που θα εκτοξεύσει το δορυφόρο. Είναι αξιόπιστος ο πύραυλος Σογιούς και οι πελάτες έχουν εμπιστοσύνη στον Σογιούς και λειτουργεί το σύστημα. Τώρα πώς καταλήξαμε να χρησιμοποιούμε τους πυράβλους Σογιούς. Ο έπρεπε να εκτοξεύσει 30 δορυφόρους περίπου. Απευθυνθήκαμε στον μόνο, ε, στη μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία που εκτοξεύει δορυφόρους από επικράτεια που ελέγχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλική Γουιάννα στην περίπτωση αυτή. Έχουμε θέματα ασφαλεία, περιορισμού που μα επευλήθησαν οι περιορισμοί από του εμπειρογνώμονε για την ασφάλεια των κρατών μελών. Ποιο είναι αυτό. Μπορείτε να το ξέρετε δορυφόρου Γαλιλαίο, αλλά μόνο από έδαφο που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο φορέα που εκτοξεύει από ελεγχόμενη επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αριάνε Πα. Η Αριάννε τότε μπορούσε να προσφέρει τρεις διαφορετικούς πυράβλους. Ένα μικρό πύραυλο των Βέγκα, αλλά δεν είναι καθόλου κατάλληλος για τις δικές μας ανάγκες. Δεύτερο πύραυλο, τον Σογιούζ. Και τρίτο πύραυλο που είναι η Αριάν 5. Το Αριάν 5, ο Αριάν 5 δεν ήταν σύμβατος για την εκτόξευση των δορυφόρων μας ε, του Γαλιλαίος. Οπότε εκ των πραγμάτων υποχρεωθήκαμε να απευθυνθούμε προς τους πυράβλους Σογιούς. Λειτουργεί καλά ο πυράβλος Σογιούς, έχει μεγάλη εξοπιστία και πουλάει τους πυράβλους η Αριάν Σπάς. Έκτοτε συνεργαστήκαμε με την Αριάν Σπάς, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και τον κατασκευαστή των Ευρωπαϊκών Πυράβλων, τον Αριάν 5, για να καταστήσουμε το σύστημα Αριάν 5 εξίσου συμβατό με τους δορυφόρους Γαλιλαίος. Τον Αύγουστο λοιπόν υπογράψαμε σύμβαση με την εταιρεία Αριάν Εσπάσου, ώστε να μας δώσει και αυτή τρεις πυράβλους Αριάν 5. Έτσι θα έχουμε ε, πλήρες το προστάσιο. Θα έχουμε τις πυράβλους Ογιούς και το Αριάν 5 για τις εκτοξεύσεις. Δεν θα ήταν καλό να θέσουμε σε τροχιά όλους τους δορυφόρους Γαλιλαίος μόνο και αποκλειστικά με τον πύραυλο Αριάν 5. Και αυτό είναι σημαντικό και για λόγους τεχνικούς. Πρέπει οι δορυφόροι να μπουν σε κάποιες τροχές και χρειαζόμαστε ευελιξία για να μπορούμε να εκτοξεύουμε όχι μόνο τέσσερις δορυφόρους κάθε φορά, αλλά και δύο δορυφόρους κάθε φορά. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και τους πυράβλους Ογιούς και τους πυράβλους Αριάν 5. Όπως είπα τώρα, ήδη ε, έχουμε ε, συμβάσεις με την Αριάνε Σπάς, σύμβαση με την Αριάνε Σπάς και έχουμε τη δυνατότητα να εκτοξεύουμε στους δορυφόρους με τέσσερις πυράβλους ε, Σογιούς και τρεις Αριάν 5. Το Δεκέμβριο θα ετοιμάσουμε νέο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, εκτοξεύσεων, να δούμε πότε θα χρησιμοποιούμε ποιον πύραυλο. Το Δεκέμβριο θα μπορούσαμε να σας δώσουμε τις πληροφορίες όσον αφορά το σχέδιο εκτοξεύσεως των δορυφόρων Γαλιλαίος. Αυτά και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Φλαμό. Ο κύριος, ε, κύριε Φακίνη έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ναι, εκείνο που θα ήθελα είναι απλά να αναφέρω το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση από την οποία προέρχομαι από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων συνδέεται όχι μόνο με το Κοπέρνικους αλλά και με την πολιτική για το διάστημα και την έρευνα και ζητούμε συγγνώμη για την απουσία του υπευθύνου. Ένα από τα σημεία που εξετάζουμε προσεκτικά αυτή τη στιγμή είναι η, η πολιτική εκτοξεύσεων για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα θέματα που προαναφέρθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Επίσης πρέπει να προσθέσω ότι με τον Κοπέρνικου στον Απρίλιο είχαμε μια πρώτη εκτόξευση και είμαστε πιο τυχεροί από τους άλλους συναδέλφους και έτσι η εκτόξευση στέφθηκε με επιτυχία. Απλά για να πω ότι αυτή η επιλογή είχε γίνει και στο τέλος τέλος μπορεί αυτό όμως να οδηγήσει στο να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν πολιτικά θέματα τα οποία θέτουν υποσυζήτηση και πάλι ποιες θα είναι οι επιλογές και το είναι ο λόγος για τον οποίο οι Sentinel-2 και Sentinel-3 που θα εκτοξευθούν κατά το 2015 ένας ε, προβλέπεται με έναν ευρωπαϊκό εκτοξευτήρα να εκτοξευθεί και ο άλλος με τον ρόκοτ. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πολιτικά ποια θα είναι τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι λύσεις που μπορεί να υιοθετηθούν. Ένα στοιχείο που επίσης πρέπει να συνεξεταστεί για τα, το Σογιούς που δεν έχει καμιά σχέση με το Κοπέρνικους ή το Γαλιλαίο είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος εκτοξευτήρας που μπορεί να εκτοξεύσει αστροναύτες που θα έχουν μετά στη συνέχεια πρόσβαση στο Διεθνή Διαστημικό ε, Σταθμό ISS είναι θέμα το οποίο λαμβάνεται υπόψη ακριβώς από τη ΣΥΠΑ και τους Ευρωπαίους να μην διακοπεί η συνεργασία με τους Ρώσους. Είναι η μόνη δυνατότητα εκτόξευσης με αυτόν τον τρόπο για το Διεθνή ε, Διαστημικό Σταθμό και επιστροφή αυτών από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πάλι στην Γη. Αυτό λοιπόν σε σχέση με τον Κοπέρνικο υπάρχουν διαφορετικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Αναφέρατε μία αλλά υπάρχουν και άλλες που πολλές από αυτές με επιτυχία και πραγματικά επίσης σε σχέση με τα δημοσιεύματα και την απήχησή τους πρέπει να πούμε ότι όλο και περισσότερο βρίσκουν την θέση τους και εντάσσονται σε αντίστοιχα δημοσιεύματα αυτές οι δράσεις. Τώρα για την κατάσταση και το θέμα το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με τον κύριο Άσμπεκ δεν είμαι σε θέση να απαντήσω για την πραγματική αυθεντική εντολή το τι προβλέπετε. Όμως ε, ο Κοπέρνικος πρέπει να είναι από πλευρά ένα εργαλείο, ένα στοιχείο ώστε να, μπορούν, να μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης και για δραστηριότητες κατά της πειρατείας θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά καθώς επίσης και για την εκφόρτωση παράνομων φορτίων ή πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων και αποβλήτων στα στη θάλασσα. Καθώς επίσης τώρα και για το θέμα των δαπανών για τις ε, διαστημικές αυτές έρευνες και εμείς ασχολούμεθα με αυτό το θέμα. Έχουμε όμως μια θετική εμπειρία σχετικά. Όταν είχαμε τη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είδαμε ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου ο αριθμός πολιτικών και δραστηριοτήτων που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αυξανόταν. Ενώ τα κονδύλια συνολικά αυτού του συνολικού προϋπολογισμού ή παρέμεναν στα ίδια επίπεδα ή συρρυκνωνόντουσαν. Αρχικά λοιπόν ο Κοπέρνικος δεν προβλεπόταν να συμπεριληφθεί στο IMFF. Ε, λόγω αυτών των αυξημένων δραστηριοτήτων και περιορισμένης χρηματοδότησης. Στο τέλος τέλος όμως, χάρη στην υποστήριξη των κρατών μελών και χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντάχθηκε ο Κοπέρνικος και τώρα κάνουμε λόγο για ένα λειτουργικό πρόγραμμα πλέον που θα λειτουργήσει σωστά και θα παράσχει τα αναγκαία στοιχεία κατά τη διάρκεια της πολιετούς δράσης του. Στο τέλος τέλος λοιπόν αυτό ήταν το σημαντικότερο σε σχέση με αυτό το στοιχείο. Πολιτική λοιπόν σπουδαιότητα. Όσον αφορά την ασφάλεια του Κοπέρνικου, όπως είπα, μία μελέτη υποεξέλιξη θα αξιολογήσει σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας αυτού του συστήματος. Δεν προβλέπουμε να υπάρξουν κάποια θέματα τα οποία θα αφορούν τις υποδομές τις ίδιες ούτε και κάποιες υπηρεσίες ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα κλιματικών αλλαγών, θαλάσσιας παρακολούθησης, ναυτικής παρακολούθησης Πρέπει να δούμε σε σχέση με τις ε, κατεπίγουσες περιπτώσεις και τις περιπτώσεις ασφάλειας ποια χρήση θα γίνει, αλλά αυτό θα αποσαφινιστεί κατά το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φακίνη. Ουσιαστικά, αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, εγώ θα ήθελα να προσθέσω και να διατυπώσω μια ερώτηση προς εμάς. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο παρακαλώ, να αποσαφηνίσετε κάπως τα θέματα έρευνας τα θέματα που αφορούν την έρευνα όσον αφορά το πρόγραμμα Κοπέρνικους και ουσιαστικά και για την συμμετοχή και τη συνεισφορά των κρατών μελών στη συμμετοχή τους όσον αφορά το ίδιο το πρόγραμμα των θεσμικών οργάνων και των ε, επιμέρους κρατών μελών σχετικά. Ευχαριστώ. Μάλιστα, απαντά ο Αρμόδιος. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Αν δούμε συνολικά όλες τις δραστηριότητες στο διάστημα όλες για τις οποίες είναι υπεύθυνε ε, και δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή και το GNSS, το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού στίγματος ε, και για τη διαστημική έρευνα, γιατί δεν μιλήσαμε πολύ για τη διαστημική έρευνα. Έχουμε 12 δισεκατομμύρια για τα επόμενα αυτά 7 χρόνια ένα μέρος αυτών συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα Horizon 2020. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια ξεχωριστή δραστηριότητα, νομίζω στο πρόγραμμα Copernicus ή GNSS, αλλά υπάρχει υποστήριξη από τον, από 2020 και υπέρ των δύο αυτών προγραμμάτων. Είναι σαφής λοιπόν εδώ η διασύνδεση σε σχέση με τους συναδέλφους μας όσον αφορά αυτό το θέμα και κατά τα άλλα όπως είπαμε είναι η ίδια Γενική Διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι λοιπόν εδώ έχουμε σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας αυτό το ζήτημα ακόμα και αν σήμερα η κατάσταση σε σχέση με το Κοπέρνικος είναι το αποτέλεσμα αυτών των διαφορετικών προγραμμάτων που συνεισέφεραν να οριμάσουν κάποια προγράμματα. Και έτσι λειτουργεί αυτό συνολικά. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τον αριθμό υπηρεσιών μελλοντικά με βάση ερευνητικές δραστηριότητες που θα συνεχιστούν στο μέλλον. Όσον αφορά τη συμμετοχή λοιπόν, είναι οι κανονισμοί και διατάξεις του ορίζοντα 2020 Horizon 2020 ε, για τα κράτη που θα συμμετάσχουν, όλα τα κράτη που έχουν ε, συγκεκριμένες συμφωνίες όσον αφορά το πλαίσιο της πολιτικής, ε, των πολιτικών για τον ορίζοντα 2020. Ταυτόχρονα για την συνιστόσα των υποδομών συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος μέχρι σήμερα. Αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον, ώστε σε σχέση με το σχεδιασμό των ε, Sentinels, των δορυφόρων που θα εκτοξεύονται και που θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα κράτη-μέλη, κατά τα επόμενα 7 έτη θα γίνει και κάποια έρευνα μέσα στο πλαίσιο μελλοντικής εποπτείας παρατήρησης της γης και στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος που δεν είναι ακριβώς ε, τα ίδια τα δικά μας κρατημέλη θα δούμε πώς μπορούν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό το σημείο εραιώνεται η συζήτηση σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν, τους επαΐοντες, τους πραγματογνώμονες για τις ε, περιεκτικές παρα, ε, παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλα τα μέλη και τα, ε, τους υπαλλήλους ότι θα έχουμε και την απογευματινή μας συνεδρίαση και θα δοθεί συνέχεια εκεί όσον αφορά τις ευρωπαϊκές δράσεις με πολύ ενδιαφέροντες εκπροσώπους ως πραγματογνώμονες. Και έτσι λοιπόν το σημερινό μας πρόγραμμα σε σχέση με τις δραστηριότητες όσον αφορά κοινοβουλευτικές επιτροπές και ε, αντιπροσωπείες είναι πολύ βέβαια στενό. Ελπίζω όμως ότι αυτό το θέμα θα μπορέσει να συζητηθεί πρωτού ε, ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.